Ja, wir haben nicht mitgeteilt, die Mitglieder, dass wir jetzt Syrien Welt Doch, doch. Haben wir extra mitgeteilt? Uh, uh, Rune, um, can you see if your coordinator, for example, comes for this uh, thing with Gilmer? Yes, but can you bit phone some well, members? you know, the minister is here. There's hardly yeah. anybody in the room. So it's a bit odd, huh? Meine και κύριοι, καλημέρα σας. σα καλοχαιρετίζω στην πρωινή μα συνεδρίαση σήμερα. Θέλουμε την οσήθιστε τακτική έκθεση της προεδρία του Συμβουλίου από πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών τη Ιρλανδία να ακούσουμε για την έκβαση του Συμβουλίου Υπουργών. Παρακαλέσαμε και τον κύριο Πιοντεμού να είναι παρόν Στόχος είναι να μπορέσουμε και την απόφαση σε σχέση με τη Συρία να συζητήσουμε. Γι' αυτό καλό είναι να μπορέσει να παραμείνει ο κύριος Ντεμόμ ένα μισά ώρα παραπάνω για να ακούσουμε να έχουμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε και τη γενική έκθεση αλλά και να συζητήσουμε συγκεκριμένα το θέμα της ε, Συρίας. Θα έχουμε και την ενημέρωση, το briefing και για το Πακιστάν σήμερα. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι λοιπόν και την δική μου έκθεση, να μην τη συζητήσουμε σήμερα για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και θέλω να πω ότι έχω τον στόχο, το σχέδιο αυτό έκθεσής μου να το αναδιατυπώσω, να το ξαναγράψω. Η απόφαση που έλαβε την Δευτέρα το βράδυ το Συμβούλιο είναι κάτι που όπως το βλέπω εγώ έχει σοβαρές συνέπειες, συνέπειες για την εργασία μας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και δεν είναι το θέμα αν είναι δυνατόν να γίνουν εξαγωγές όπλων ή όχι στη Συρία. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα. Εγώ είμαι κατά των εξαγωγών όπλων, γιατί δεν ξέρουμε στο τέλο τέλο, αν μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποιο είναι τελικός χρήστη από τέτοια όπλα που εξάγονται και το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα ίσως και εναντίον μας. Όλα τα παραδείγματα δεν είναι βέβαια απόλυτα σωστά, αλλά οι Αμερικανοί πρώτα εξόπλισαν τους Ταλιμπάν κατά των Ρώσων και μετά οι Ταλιμπάν χρησιμοποίησαν αυτό, αυτά τα όπλα, ε, στράφηκαν εναντίον μας. Μετά εξόπλισαν τον Σαντάμ Χουσεΐν ε, οι Αμερικανοί, αυτός πήγε όμως και εισέβαλε στο Χουβέιτ μετά. Και στο τέλος τέλος ε, πρέπει να δούμε όχι μόνο το θέμα του Ασάντα, αλλά μήπως έρθουν οι ακραίοι Ισλαμιστές στην εξουσία στη Συρία που δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκεί με κάτι τέτοιο και θα αρχίσει το κυνήγι κατά των μειονοτήτων. Και σε σχέση με, τους, ε, με τον φονταμεταλισμό δεν θα πρέπει να πει κανείς ότι υπάρχουν ε, μόνο απλά και κάποιοι άλλοι φιλελεύθεροι, πιο φιλελεύθεροι ε, μουσουλμάνοι Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όλες αυτή η απόφαση έχει επί των αρχών σημαντικές επιπτώσεις. Η απόφαση σημαίνει ότι σκιαγραφείται ότι δεν θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον αρμοδιότητες για τα θέματα εξαγωγής όπλων ως Ένωση. Και ότι όλα αυτά επανεθνικοποιούνται πλέον ξανά, επανεθνικοποιήθηκαν. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν για τους Βρετανούς αυτός ήταν ο κυριότερος στόχος και όχι ο κυριότερος στόχος η Συρία π.χ διότι όταν λένε ότι τους επόμενους δύο μήνες δεν θέλουν να δώσουν όπλα, ε, τότε θα μπορούσαν να είχαν δεχτεί τον συμβιβασμό που προέβλεπε κάτι τέτοιο, δηλαδή την απόφαση μετά την Σύνοδο της Γενέβης 2. Επί της δεν είναι τίποτα διαφορετικό, είναι όμως η αφαίρεση της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας για τα θέματα εξαγών όπλων και επανεθνικοποιείται το θέμα. Και αυτή η επανεθνικοποίηση έχει βαθύτατες επιπτώσεις που πρέπει να τις δούμε και να τις λάβουμε υπόψη. Εδώ προτάσεις ε, πανεθνικοποίησης, ε, η ένταξη στις εθνικές αρμοδιότητες από πλευράς ε, των Βρετανών με εξαιρετική χρήση εκμετάλλευσης του δικαιώματος αρνησικηρίας καταλήξαν στο να επιτευχθεί εν μέρει αυτός ο στόχος. Και θα λέγα ότι κάποιοι δεν το είχαν συνειδητοποιήσει αυτό την νύχτα της Δευτέρας. Ο κύριος Χέιγκ είπε στην αρχή της συνεδρίασης ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή πολιτική αλλά για βρετανικά συμφέροντα μέσα σε ένα πλέγμα. Δηλαδή καθορίζει το θέμα με καθαρά εθνικούς όρους, με όρους παιχνιδιού εθνικής πολιτικής. Και αυτό ως θέμα αρχής. Μπορεί να τον συγχαρεί κανείς βέβαια για αυτό πόσο, με πόσο ευφυή τρόπο τα κατάφερε και τα πέτυχε αυτά που ήθελε να πετύχει. Οι Βρετανοί δεν χρειάζονται πια δημοψήφισμα, μια και σε σχέση με τη διαπραγμάτευση αρμοδιοτήτων, με γεγονότα αυτού του είδους, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, με κοινικό τρόπο, κατάφεραν το στόχο τους. Αλλά φτάνουν τώρα τα εισαγωγικά οι παρατηρήσεις μου. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Thank you, uh, uh, Chairman, and uh, thank you again for the opportunity uh, to be. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να είμαι σήμερα εδώ. Για να είμαι σύντομος, ε, θα μιλήσω για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Μαΐου. Η Σύνοδο του Συμβουλίου, όπως είπατε, αφοσιώθηκε κυρίως το θέμα της Συρίας και την απόφαση για το μέλλον των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το εμπάργκο για την πολυσιόπλων, στο οποίο θα επανέλθω εντό ολίγου. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη έχουν την κοινή πεποίθηση ότι έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξευρεθεί πολιτική λύση και πρέπει να γίνει αυτό για να δοθεί τέλος στην σύγκρουση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει τη στήριξή της προς την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ώστε οι πλευρές να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βάσει του ανακοινοθέντος της Γενέβης του Ιουνίου 2012. Όπω τονίζουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται για να βρεθεί λύση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τον Σύνδεσμο Αραβικών Εθνών, τον κύριο Μπραχήμη και τον ε, Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τα συμπεράσματα καλούν την αντιπολίτευση του Σταυρισμού της Συρίας και όλα τα πολιτικά, τις πολιτικές ομάδες να αναζητήσουν πολιτική λύση της διαμάχης και να ειρηνεύσει η χώρα. Οι ανθρωπιστικές ε, διαστάσεις της καταστροφής ε, αντικατοπίζονται επίσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου διότι 80.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1,5 εκατομμύριο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η κλίμακα της καταστροφής παίρνει όλα ένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα μέλη θα γνωρίζουν ότι υπάρχει ουσιώδης στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη με πάνω από 700, 700 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ που έχουν εκταμιευθεί και άλλα που πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσφατα. Οι Υπουργοί δεσμεύτηκαν για 12 μήνες να λάβουν δεσμευτικά μέτρα για το εμπάργκο όπλων. Και όπως συμφωνήθηκε, υπάρχει μια δήλωση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου με δέσμευση των 100 μελών να τηρήσουν μια σειρά από εχέγγυα μέσω της διεθνή πολιτικής ως προς την ε, προσφορά στρατιωτικού υλικού. Η δήλωση τονίζει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα προχωρήσουν σε αυτή τη φάση στην ε, προσφορά ή οδήποτε εξοπλισμού εντό διμήνου. Η θέση αυτή θα επανεξεταστεί βάσει τη έκθεση τη τη εκπροσώπου για τι πρόσφατε εξελίξει. Κυρίω ε, θα εξαρτηθούν όλα από το κατά πόσο οι διαφορετικέ πλευρέ θα συμμετάσχουν στη διαδικασία τη Γενέβη και θα φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ύπατη εκπρόσωπο θα συζητήσει επίση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πριν υποβάλει την έκθεσή τη. Η ανταλλαγή απόψεων για την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή είναι κάτι που αναμένεται αλλά δεν έχει προχωρήσει λόγω χρονικών περιορισμών. Θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για να δούμε πώ προχωρούν οι αμερικανικέ προσπάθειε, να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο πλευρών, να βρεθεί μια λύση και να αρχιστεί το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Ε, σω αυτή να είναι και καλύτερη ευκαιρία για να δούμε κατά πόσον υλοποιήθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το Μάιο και το Δεκέμβριο τη περασμένη χρονιά η ένταση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζεται το γεγονό ότι οκτώ ε, Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επισκεφθεί την περιοχή από τον, τη Σύνοδο Συμβουλίου του Απριλίου και μετά. Επίση, το ε, Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων συζήτησε και για την πολιτική ασφάλεια και άμυνα, ε, όπου οι Υπουργοί εξέφρασαν τι απόψει του εν ώψη τη ολοκλήρωση τη έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη ΕΠΑ εκπροσώπου και βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο και των συζητήσεων των Υπουργών να μείνει τον Απρίλιο. Εδώ δόθηκε προσοχή στην διαχείριση κρίσεων ε, για τους πολίτες και αυτό ήταν ένα θέμα που ως τώρα δεν είχε λάβει τόσο μεγάλη διάσταση εν ώψη Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, οργανώθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση πολιτικών κρίσεων, συγκεκριμένοι στόχοι για τις αποστολές ε, πολιτικής προστασίας, συγκεκριμένες στρατηγικές και οι συσχετισμοί μεταξύ της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και άλλων πολιτικών, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η αναθεώρηση της πολιτικής αυτής θα βοηθήσει στην ε, πρόθεση της. Η... Είπατε εκπρόσωπο τη εισαγωγική τη παρατηρήση έθιξε αρκετά θέματα που θα περιέχονται και στην έκθεση. Αναφέρθηκε στο επιτυχέ αποτέλεσμα τη ε, Συνόδου των Δωρητών στο Μαλί για το Μαλί μάλλον, που οργανώθηκε το Μάιο στις Βρυξέλλες. 108 αντιπροσωπείες συμμετείχαν, ε, πολλοί επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων και υπουργοί εξωτερικών μεταξύ τους. Το συνολικό ποσό που θα δεσμευτεί έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες με περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 120 εκατομμύρια ευρώ. Ε, θα δοθεί ε, προσοχή στην υλοποίηση των υποσχέσεων και του σχεδίου ανάκαμψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκταμιεύσει κονδύλια για το Μαλί και έχει δεσμευτεί να κάνει σχετικά προτάσει. Το Συμβόλαιο εφέτησε τα συμπεράσματα, τονίζοντα τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση του μεταβατικού οδικού χάρτη, βάσει τη απόφαση τη εκπροσώπου να υπάρξει και ε, παρατήρηση των εκλογών και σχετική αντιπροσωπεία για παρατήρηση των εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, ο διαρθρωμένος διάλογο με το Βελιγράδι και την Πρίστινα είναι ένα θέμα στο οποίο ε, μας ε, σταθήκαμε και δεσμεύτηκε και σε αυτό είπατε εκπρόσωπο να επιτελεστεί πρόοδος. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο τη χρονιά, με την ανάληψη δράση ήδη από την επόμενη εβδομάδα για θέματα όπω ο νόμο περί αμνηστίας και η τόνωση των υποδομών του δικαστικού και αστυνομικού κλάδου. Τώρα, για τη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Σομαλίας στις 16 Σεπτεμβρίου ε, υπάρχει ήδη προετοιμασία με δύο συναντήσεις ήδη την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει στρατηγικό πρόγραμμα για να ανασυσταθεί το κράτος αυτό και να μελετηθεί η προσχώρηση της Σομαλίας στην Συμφωνία Κοτονού μέχρι το Σεπτέμβριο. Πρόεδρε, με τα χαράς να απαντήσω σε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής σας. Κύριο Σαλαφράγκα, σα ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα το πρωί να μας πληροφορήσετε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων αυτής της εβδομάδας. Θα ήθελα να σας πω σε σχέση με τη Συρία ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι σημειώνουμε τις πολιτικές των κρατών μελών για τις εξαγωγές όπλων και αυτές λαμβάνουμε υπόψη, δεν θα εγγραφούν στα Μητρώα και στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν μια από τις πιο ένδοξες συνέπειες και ένα από τα πιο ένδοξα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών και χωρίς αναφορά σε σχέση με την επανεθνικοποίηση όπως είπε ο πρόεδρος ε, των κοινοτικών αρμοδιοτήτων ή την επιβολή της θέσης ενός κράτους μέλους σε σχέση με τον προσανατολισμό στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα είναι ένα θέμα πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σπουδαίο σε σχέση με την απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Συρία και είναι προφανές ότι το Συμβούλιο Υπουργών είχε διχαστεί σε βάθος, είχε βαθιά διχαστεί και είναι επίσης σαφές ότι συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Στα, στο 3 δεν είναι γαλλικά που ακούγονται αλλά σλοβενικά έρχονται στο κανάλι 3 που είναι το κανάλι των γαλλικών. Αυτό σε σχέση με τους διερμηνείς να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει κύριε Σαλαφράγκα. Έλεγα δεν αναφερόμουν τόσο στην σπουδαιότητα που μπορεί να έχει η επανεθνικοποίηση μιας κοινοτικής πολιτικής όπως είναι μια εμπορική πολιτική ούτε στην επιβολή των κριτηρίων για τον προσανατολισμό στο Συμβούλιο των απόψεων ενός κράτους μέλους, αλλά περισσότερο για την θλιβερή, πολύ σημαντική απώλεια ζώων στην ε, Συρία και όπως ε, και το Κοινοβούλιο στην, ε, στο ψήφισμά του σε σχέση με αυτό το θέμα στην προηγούμενη Ολομέλεια και όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Επίσης θα ήθελα να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων προσπαθώντας να εντάξει τις διάφορες εναλλακτικέ δυνατότητες σε σχέση με το Συμβούλιο των Υπουργών όσον αφορά τον αποκλεισμό, το εμπάργο για την εξαγωγή όπλων στη Συρία. Αλλά εμένω και επιμένω το ότι το να λάβουμε υπόψη είναι αυτό, αυτή την κατάσταση σε σχέση με τις θέσεις των κρατών μελών, εδώ πρέπει να διατυπωθεί ένα ερώτημα, Πρόεδρε. Και με τα επιχειρήματα, χωρίς να πέσουμε σε ένα υπερβολικό δραματισμό, υπερδραματικοποίησης ε, της κατάστασης, πρέπει να διαρωτηθούμε πόσοι περισσότεροι θάνατοι θα προκληθούν. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αυτούς τους δύο μήνες είχαμε τρομερή απώλεια ζώων ε, στη Συρία και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, για να φτάσουμε στο σημείο να σημειώνουμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις ατομικές πολιτικές των κρατών μελών, γιατί αναμείναμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί περιμέναμε δύο ολόκληρα χρόνια να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που ίσως θα μπορούσαν να είχαν σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές, αν δεν είχαμε καθυστερήσει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανα, ανα, ανα, η κυρία Γκόμες, πρόεδρε, ο κύριος Σαλαφράγκα ήταν πολύ διπλωματικός στις αναφορές του. Ε, και εγώ είμαι εξ επαγγέλματος ε, διπλωμάτης. Αλλά η επανεθνικοποίηση των εξαγωγών όπλων είναι κάτι που το χαρακτήρισε ως ε, πολύ κακή εξέλιξη και δεν θα πω περαιτέρω, δεν θα κάνω σχολιάσω περαιτέρω. Γιατί είμαι βέβαιη ότι θα τοποθετηθεί σχετικά το Κοινοβούλιο. Μιλάμε για εξαγωγές όπλων. Μιλάμε για όπλα που σε πολλά μέρη του κόσμου είναι όπλα μαζικής καταστροφής. Σε ό,τι αφορά τη Συρία, να ρωτήσω το εξής. Το Συμβούλιο σκέφτηκε να δημιουργήσει κάτι τόσο θεμελιώδες όπως μια ομάδα επαφής στα πλαίσια του ΟΗΕ, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Δηλαδή η Ρωσία και η Κίνα κυρίως. Και όχι απλώς για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά για να υπάρχει κοινή ανάληψη ευθύνης. Αυτό Το είδαμε και σε προηγούμενα παραδείγματα και είναι κάτι που έχουμε μάθει από το παρελθόν, από τα Βαλκάνια λόγω χάρη. Γιατί δεν γίνεται για τη Συρία. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω εάν σκέφτηκε ε, το Συμβούλιο τρόπους να να δει τι γίνεται με τους διάφορους, ε, διάφορες πλευρές που έχουν ε, συσπηρωθεί σε διαφορετικά σημεία της χώρας, της ε, επικράτειας της Συρίας, πώς μπορούν να οργανωθούν και να περάσουν σε διάλογο. Νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τα βασικά τα θεμελιώδη που θα πρέπει να έχουμε διδαχθεί από άλλες κρίσεις. Και αυτή η συγκεκριμένη κρίση είναι προφανώς πολύ σοβαρότερη από πολλές οπτικέ γωνίες λόγω της ριζοστη... ριζοσπαστικοποίησης ε, στο... στο κέντρο της Μέσης Ανατολής. Επίσης, με ενδιαφέρει τι συζητήσεις έγιναν γιατί το επόμενο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα ασχοληθεί και με μια θαλάσσια στρατηγική ασφαλείας θα υπάρξει συνεννόηση με τους ε, υπουργού αμήνης ή αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τους υπουργού αμήνας ή θάλασσα, θεωρείται επικάλυψη προσπαθειών, δεν τους νοιάζει. Ο κύριος Λάμπστορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μόλις τώρα είπε η κυρία Γκόζμες ε, Πράγματι αυτή ήταν μια ε, επονίδιστη ημέρα για την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής ημέρας. Πριν από τη συνάντηση οι υπουργοί από διάφορες χώρες είχαν εμφανιστεί στην τηλεόραση και είχαν δηλώσει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ενωσιακή ενότητα για να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ε, στη διεθνή αρένα. Διαπιστώσαμε όμως ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αν οι ίδιοι υπουργοί δεν την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Ο πρόεδρος ε, υπενήχθη τη θέση των Βρετανών, η οποία όμως ήταν ξεκάθαρη ευθύς εξ αρχής. Το Λονδίνο δεν ήθελε να συνεχιστεί το εμπάργο και ε, επειδή ε, υπάρχει, προβλέπεται ομοφωνία για τέτοιου είδου θέματα, αυτό είναι λάθος στη συνθήκη, η Μεγάλη Βρετανία κατόρθωσε τελικά να επιβάλλει τη δική της τη βούληση σε όλους τους άλλους. Η Γαλλία συμφώνησε με τη Βρετανία αλλά αυτό μοιάζει να είναι ένα μοντέλο της ε, ευρωπαϊκής ε, κακοδαιμονίας. Ε, κάποιες χώρες όταν τις βολεύει, συμπεριλαμβανομένες και τις δικής μου, συνεργάζονται με τους Βρετανούς. Όταν ε, πρόκειται ας πούμε για περικοπές στον προπλογισμό, η Γερμανία με χαρά τη συνεργάζεται με τη Μεγάλη Βρετανία και όλοι οι άλλοι τις ανασχετούν. Γίνεται όμως αυτό. Οποτεδήποτε πρόκειται για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Γαλλία ε, συνεργάζεται με τη Βρετανία. Δεν τα λέω όλα αυτά ε, με κοινικό ύφος, απλά είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον εαυτό της. Επίσης, πιστεύω ότι η θέση των ε, Βρετανών προφανώς ή είναι δυνατόν να διαμορφώθηκε από τα συμφέροντά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα συμφέροντα των Βρετανών δεν νομίζω ότι διαφέρουν ουσιαστικά από τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σε τελική ανάλυση δεν ενδιαφέρει όλους μας να εξευρεθεί μια πολιτική λύση, μια διαδικασία που θα εμπορίσει ή θα εμποδίσει η κρίση αυτή να μεταπηδήσει σε γειτονικέ χώρες, ε, στην Τουρκία. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν συμπίπτουν με τα βρετανικά. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω από εσά, κύριε Υπουργέ, ε, ποια ε, συμφέροντα δήλωσε η βρετανική πλευρά που κατά την άποψή της ε, διαφέρουν από τα ευρωπαϊκά έτσι ώστε τελικά να μην υπάρχει ενότητα. Πρόεδρε, αυτό δεν συμβαίνει ούτε πρώτη φορά, ούτε δεύτερη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει λόγω ε, εθνικών συμφερόντων. Η πρώτη ήταν η Λιβύη. Εκεί η Γαλλία ε, προπορεύτηκε στο Μαλί επίσης ε, και τώρα είναι η τρίτη φορά στην Συρία η Βρετανία και η Γαλλία σπάνε την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Εγώ προτείνω να διαγράψουμε αυτά που ελέγξαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Από ό,τι φαίνεται ήταν όλα περιτά. Εάν λοιπόν οι αρχηγοί ε, κρατών και κυβερνήσεων επιθυμούν να δαπανούν, να σπαταλούν τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, ε, δικαίωμά του να το κάνουν, αλλά ε, τουλάχιστον θα έπρεπε να το σκεφτούν σοβαρά. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω ότι όλοι οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν με θέματα περιεχομένου και μορφής και πρέπει να πω ότι η απόφαση που ελήφθη ήταν η χείριστη δυνατή. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η συλλογιστική άρση στο εμπάργκο των, της πώληση όπλων, εκτός και αν πρόκειται για ένα ημίμετρο για να καθησυχάσουμε τις συνειδήσεις μας. Δεν μπορεί η άρση του εμπάργου πώληση όπλων ήδη με τη διαδικασία που προβλέπεται να υλοποιηθεί με προθεσμίες, με μήμετρα, με συγκεκριμένε ημερομηνίε να κάνει κάποια σοβαρή διαφορά στην πράξη. Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Η εναλλακτική είναι σαφής. Είτε θα έχουμε στρατιωτική παρέμβαση και μάλιστα η στρατιωτική παρέμβαση για να σταματήσει σφαγή είτε θα ξέρουμε μια πολιτική λύση. Η λύση που έχει προταθεί τώρα είναι φρικτή, αποτρόπαιη από ηθικής άποψη σε σχέση με αυτά που βλέπουμε να γίνονται καθημερινά. Και από διεθνού διπλωματική άποψη βλέπουμε οτι έχει γίνει με άλλες συγκρούσει και σειράξει. Στα Βαλκάνια λόγου χάρη, ξέραμε τι συνέβαινε στην Βοσνία, εκεί ε, είδαμε καθημερινέ σφαγέ και η πολιτική ήταν lift and strike τότε. Το σημαντικό όμω και εκεί που δόθηκε έμφαση ήταν στο χτύπημα, το στρατιωτικό χτύπημα. Πώ γίνεται να έρθει το εμπάργκο χωρί να υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση και ούτε διπλωματικέ συνομιλίε. Είναι απολύτω περιττό, θα ενισχύσουμε απλώ τη σύγκρουση και θα έχει τεράστιε συνέπειε αυτό, φρικτέ και σε εμά του ίδιου. Στο Λίβανο, στα υψίπεδα του και ούτω καθεξής. Θα προτιμούσα λοιπόν το Συμβούλιο να αξιοποιήσει το δεκάωρο συζητήσεων και να συζητήσει για τη διάσκεψη της Γενέβης έστω και την περίφημη πολιτική μάλλον λύση την οποία όλοι στηρίζουμε εδώ και μήνες. Εδώ δεν έγινε τίποτα και δεν έχουμε ευρωπαϊκή απάντηση στα αυτά τα θέματα. Θα συζητήσουμε με τον Ασάντ, διότι αν θέλουμε πολιτική λύση πρέπει να συζητήσουμε με όλους. Θα έρθει το Ιράν, Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα. Αυτά τίθενται σήμερα και θα υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος της ε, διαπραγματεύσεις. 11 ώρες ε, συζητήσεις για ε, νομικίστικους γρίφους για να δούμε πώς θα καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας χωρίς να πληρώσουμε και τίποτα. Για την εξωτερική μας εικόνα δηλαδή. Το βρίσκω πραγματικά θλιβερό όλο αυτό. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ομιλώ εκ μέρου ε, τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά τυχαίνει να ανήκω ε, σε ένα από τα κόμματα ή στο κόμμα, το οποίο επίση συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού. Και με κάθε σεβασμό ε, στου άλλου συναδέλφου, κυρίω προ τον κύριο Λάμπστορφ, πρέπει να σα πω ότι δεν ήταν λάθο τη συνθήκη τη Λισαβόνα να προβλέπει την ομοφωνία στην εξωτερική πολιτική, που θεωρείται το προπύργιο τη Ευρωπαϊκή Ενότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλες σημαντικές χώρες θα το, έβρεπαν, θα το θεωρούσαν αδύνατον, απαράδεκτο να μπορούν άλλες χώρες μικρότερες ίσως να ανατρέψουν την ε, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να αρθεί το εμπράγκο. Το είχε πει και παλαιότερα μετά από ε, πραγματικά στάθμιση των κινδύνων και στόχος δεν ήταν ε, βέβαια να προκληθεί περαιτέρω αιματοχυσία ή να ε, διχαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς στόχος ήταν ε, η κυβέρνηση Ασάντ να μην μπορεί να προβεί και σε περαιτέρω σφαγές, να σταματήσει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Το Ιράν, η Ρωσία, η Κίνα και η Χεσμολά όλο και περισσότερο με πολλούς στρατιώτες παρόντες στη Συρία μάχονται και επίσης ε, και μία παρένθεση πρέπει να δούμε και τι γίνεται τελικά και με τον κατάλογο τρομοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όλα σε σχέση με τον Ασάντ και με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε δυστυχώς να εξοπλίσει τους ε, μετριοπαθείς ε, αντιστασιακούς. Απευθύνομαι στον Ζελί Μεντρίς ε, που είναι ο αρχηγός του Ελεύθερου Στρατού της Συρίας. Μου φάνηκε μετριοπαθής άνθρωπος και δυστυχώς αυτός δεν μπορεί να εξοπλιστεί. Ίσως θα πρέπει να του εξοπλιστούν, μετά βέβαια να παρακολουθείτε η όλη κατάσταση από ειδικού ε, παρατηρητές. Ε, ίσως λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί επιτάπητος ε, στη συνάντηση για τη Γενέβη που θα λάβει η χώρα. Γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι οι σαλαφιστές και η Αλκάιντα αν, πάρουν, αν αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα όπλα αυτό θα είναι τραγικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να αστυνομεύουμε την κατάσταση επιτόπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, θα μιλήσω γερμανικά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εκπλήσει το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω, εγώ δεν εκπλήσωμαι, απλά λαμβάνω υπόψη μου ε, το ε, τι ακριβώς ε, αποφάσισε το Συμβούλιο σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν οδηγεί σε κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά τελικά αφήνει τη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όταν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή άποψη για τέτοιου θέματα, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Βεβαίως μπορεί να διήστανται απόψεις ε, για το ποια μπορεί να είναι η ΚΕΠΑ. Εμείς λέμε προφανώς ε, δεν επιθυμούμε στρατιωτικές λύσεις. Εδώ όμως αποδεικνύεται η αδυναμία να ε, καταλήξει κανείς στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους συγκρούσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίδραση της κοινή γνώμης. Επιπλέον, θεωρώ ότι αν το Συμβούλιο το Κοινό Συμβούλιο βάλει την κοινή εξωτερική πολιτική ε, ως ένα βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, τότε θα πρέπει ε, και η ύπατη εκπρόσωπος ε, να εξηγήσει, να παρουσιάσει την εξέλιξη της κοινή θέση. Οι πολίτες ε, σε όλα τα κρατημέλη πρέπει να μπορούν να διαπιστώσουν πώς επιθυμούμε να χαράξουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, ε, λόγω της ε, πραγματικότητας στα κράτη-μέλη θα προκύψουν συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών, κάτι που δεν εξυπηρετεί κανένα, δεν ε, στηρίζει ούτε την διεθνή εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω και μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί τελικά δεν προέκυψε σαφέστερη θέση όσον αφορά το πρόβλημα των προσφύγων. Ο κύριος Αλαφράνκα μέχρι τώρα ήταν ο μόνος που επισήμανε την ανθρώπινη διάσταση στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουμε ευθύνη πρέπει να υπάρξουν σαφέστερες απόψεις όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων. Εγώ τουλάχιστον αυτό περίμενα και σας μπορείτε να ε, τοποθετηθείτε περαιτέρω επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ως προς την ε, διάσταση του προβλήματος, την εμβέλεια που έχει λάβει η κατάσταση της Συρίας. Με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις, 80.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν από τη χώρα. Πρόσφυγες στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Πάνω από 6 εκατομμύρια χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμη και τη στιγμή που αρχίσαμε να συζητάμε σήμερα το πρωί, πόσοι θανατώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους στη Συρία. Πόσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και τις αιστείες τους. Με ένα τέτοιο σκηνικό, νομίζω ο κύριος Νταζό το έθεσε έτσι. Πώς οφείλουμε να αποκριθούμε στην κρίση αυτή. Στρατιωτική παρέμβαση χρειάζεται, όποιας μορφής και αν είναι, για να σταματήσει ο σφαγιασμός. ή θα πρέπει να εξεύρουμε μια διπλωματική πολιτική λύση. Η στάση που αποφάσισε να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση είναι να ακολουθήσει ειρηνική πολιτική διπλωματική οδό και διευθέτηση του προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς στηρίζει τη διαδικασία Μπραχήμη και όσα προβλέπει αυτή η ευρωπαικη ενωση διαρκως στηριζει τη διαδικασια εμπραχημη και οσα προβλεπει αυτη η διαδικασια και γι' αυτό ακριβώς συμφωνούμε βάσει των συμπερισμάτων του Συμβουλίου της Δευτέρας, συμφωνούμε με την πρωτοβουλία Πολιτείων και Κίνας και την έναρξη της λεγόμενης διαδικασίας Γενέβη 2. Αυτό που ακούστηκε από την κυρία Γκόμες, δηλαδή γιατί δεν υπάρχει ομάδα επαφής στη διαδικασία της Γενέβης προβλεπόταν μια ομάδα δράσης. Συμμετείχαν 10 χώρες, συν ε, επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή άρχισε να λειτουργεί ως μέρος της διαδικασίας Γενέβη 2. Η ύπατη εκπρόσωπος βρίσκεται σε διαρκές επαφέ με τους ε, εμπλεκόμενους στην σύραξη και τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος φορέας ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και προσφέρει ανακούφιση στους πρόσφυγες. Αυτό είναι κάτι που έθεσε ο κύριος Σόλτς σε σχέση με την κατάσταση των προσφύγων, την ανθρωπιστική τους κατάσταση και είναι και κάτι που ρητός ε, σχολιάζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η ενασχόλησή μας με τη Συρία δεν ε, ασχολείται αποκλειστικά με την άρση του εμπάργου. Υπάρχουν τρεις σελίδες και μια σειρά από συμπεράσματα που αφορούν τη Συρία και συγκεκριμένα αφορούν την ανθρωπιστική διάσταση του θέματος, το τι γίνεται με τους πρόσφυγες και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τη σχετική κατάσταση. 100 ε, εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται με 700 ήδη να έχουν εκταμιευθεί. Τώρα για την άρση του εμπάργου. Όπως είπε ο κύριος Λάμστορφ, η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί ομόφωνα. Αυτό που συζήτησε όμως το Συμβούλιο τη Δευτέρα ήταν η επανάληψη των κυρώσεων. Το καθεστώς των κυρώσεων, δηλαδή το εμπάργκο συμπεριλαμβανόμενο, πνέει στο τέλος του μήνα, εκτός και αν ανανεωθεί, αν αποφασιστεί να ανανεωθεί. Το καθεστώς κυρώσεων συμπεριλαμβανομένου του εμπάργου όπλων απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για να ανανεωθεί. Υπήρξε ομοφωνία εν τέλει για την ανανέωση των κυρώσεων, των οικονομικών, των εμπορικών, των ε, δημοσιονομικών και ούτω καθεξής. Τα μέτρα δηλαδή, τα κατασταλτικά. Αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία, δεν υπήρξε ομοφωνία για την ανανέωση του εμπάργου όπλων. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναζητήσει μια συμβαστική λύση για την διόρθωση του εμπάργου ή θα μπορούσε απλώς να έχει διαφωνήσει για την ανανέωση του εμπάργου όπλου. Οπότε μετά περνάει το θέμα στα χέρια των επιμέρους κρατών μελών να αποφασίσουν πώς θα δράσουν. Αντί να μείνει το θέμα ανοιχτό, συμφωνήθηκε να υπάρξει αυτή η δήλωση, στην οποία προσχώρησαν όλα τα κράτη-μέλη, προσυπέγραψαν μάλλον όλα τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να ε, καταγράψουν μια σειρά από προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για την ε, προμήθεια όπλων. Λόγου χάρη, η παράδοση όπλων θα γίνεται μόνο προς τον Εθνικό Στατό της Συρίας. Δεν πρόκειται για παροχή όπλων γενικώ και ορίστος. Αυτό είναι κάτι που τόνισαν πολλά από τα μέλη της Επιτροπής σας το κατά πόσον δηλαδή μπορούμε να παρακολουθούμε πού θα καταλήξουν τα όπλα, σκοπός είναι να προστατευτούν οι άμαχοι. Θα απαιτηθούν βέβαια και έχει έγκυα για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να, αποτιμήσουν το πώς εφαρμόζονται οι εξαγωγές τους αδειοδοτήσεις και βάσει των κριτηρίων που έχουν προκύψει από την κοινή θέση του Συμβουλίου από τις 8 Δεκεμβρίου Σεπτεμβρίου του 2008 που καθορίζει κοινού κανόνε που διέπουν την εξαγωγή αισθητικού εξοπλισμού με πολύ συγκεκριμένε ε, και αυστηρέ αρχέ. Τέλο, συμφωνήθηκε τα κράτη-μέλη να μην προχωρήσουν σε αυτή τη φάση με την παροχή εξοπλισμού. Εγώ αυτήν την δέσμευση την ερμηνεύω όχι χρονικά, ως χρονική περίοδο όπως ε, δημοσίως ερμηνεύτηκε, δεν μιλάμε δηλαδή για την ημερομηνία στην οποία το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τη θέση του και θα αντιστραφεί η κατάσταση. Όχι. Θέλουμε απλώ η διαδικασία τη Γενέβη να προχωρήσει εντωμεταξύ και εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την τοποθέτηση αυτή του Συμβουλίου. Νομίζω, για να είμαστε δίκαιοι και επειδή έγινε πραγματικά εντατική συζήτηση, κανείς δεν πρόβαλε στη συζήτηση αυτή τα δικά του εθνικά συμφέροντα. Η συζήτηση περισσότερο πραγματικά κατέβαλε ουσιαστικέ προσπάθειες να βρεθεί μια αληθινή λύση. Κανείς δεν επεδίωξε τα δικά του ατομικά συμφέροντα εντό εισαγωγικών στη συγκεκριμένη συζήτηση. Αυτό που ακούστηκε ως ε, άποψη είναι ότι έπρεπε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Δυστυχώς δεν υπήρξε ομοφωνία για την ανανέωση του εμπάργου όπλων. Οπότε αυτό που πια έχουμε στα χέρια μας είναι ισχυρά πολιτικά συμπεράσματα μεν για τη Συρία, όπου καταγράφεται η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαδικασία εξέβρεσης λύσης, ως προς την ανθρωπιστική επίγουσα κατάσταση και από την άλλη υπάρχει και η δήλωση για την άρση των εμπαργόπλων. Απλά επειδή αρκετοί ομιλητής μίλησαν για τα θέματα τη ε, ΚΕΠΑ. Η συζήτηση για τα θέματα ΚΕΠΑ ήταν μια προπαρασκευή για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Είναι μία από πολλές συζητήσεις που διεξάγονται και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στις συναντήσεις των Υπουργών Άμυνας. Θα υπάρξουν άλλες τέτοιες συζητήσεις πριν από το Συμβούλιο Δεκεμβρίου η ειδική ιδιαίτερη συζήτηση που είχαμε σε σχέση με τη Δευτέρα επικεντρωθήκε στην πολιτική πλευρά της ε, ΚΕΠΑ. Αλλά όπως είπα είναι μία από πολλές ε, περισσότερες συζητήσεις που διεξάγονται σε σχέση με το ζήτημα αυτό και ειδικότερα στο θέμα της ε, ναυτικής, ναυτιλιακής πολιτικής που φυσικά είναι ένα σημαντικό μέρος στην εξίσωση αυτή δεν επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα σε αυτό το Συμβούλιο αυτού του μήνα Υπουργών Εξωτερικών, αλλά αναμένω ότι θα υπάρξουν και άλλες ε, ευκαιρίες όπου θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Κύριος Πανσέρη, uh, παρακαλώ, έχει τον λόγο, εντάξει. have asked about... Τα εσείς. Yeah, that wasn't discussed on Monday. Για τη Χεσμολά δεν συζητήσαμε, δεν είπαμε τίποτα τη Δευτέρα. Ο κύριος Παντσέρη παρακαλώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ δεν θα είμαι και τόσο διπλωματικός. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Σαλαφράγκα που είπε ότι η απόφαση που έλαβε το συμβίλιο δεν είναι και καμιά φοβερή απόφαση δεν είναι για να χαιρόμαστε. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι τελικά ε, προβλήθηκε η πολιτική υποκρισία, το εμπάργκο δεν θα εννοηθεί και τελικά κάθε χώρα θα κάνει αυτό που θέλει. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την Ευρώπη έχουμε πλέον ε, περάσει στο δυνατότητα αυτοεξαίρεση σε κοινωνικές, κοινωνικές πολιτικές αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Εσείς λέτε ότι κανείς δεν θα στείλει τελικά όπλα μέχρι νεοτέρας ε, ε, και θα πρέπει να ελέγχουμε τι θα γίνεται επί Όσον αφορά το θέμα των όπλων, υπάρχει το πρόβλημα μήπως τα όπλα αυτά πέσουν στα χέρια τρομοκρατών. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθούμε τη διαφωνία να την καλύψουμε με ένα φύλλο Ο κύριος Υπουργό θα πρέπει να ξέρει ότι η απόφαση του Συμβουλίου προκάλεσε ήδη την απόφαση της Ρωσίας ε, που είπε ότι θα του στείλει του Ασάτ ε, τα S300 τους πυράβλους ε, σε τρακόσια... Και αυτό βέβαια προκάλεσε αντίδραση ε, από το Ισραήλ στον Υπουργό Άμυνας. Πρέπει να προσθέσουμε και την εκρηκτική κατάσταση των προσφύγων. Νομίζω λοιπόν, μπράβο σας, συγχαρητήρια, αριστούργημα αυτό, αυτή η απόφαση της εξωτερικής πολιτικής ε, για την ε, διαφύλαξη της ειρήνης. Τα τελευταία, τις τελευταίες ώρες είδαμε ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση η κούρσα των εξοπλισμών μπορεί τελικά να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες. Λοιπόν, λοιπόν την εντύπωση ότι αντί να περνάμε ε, τον ώρα μας ε, δίνοντας ε, δίθεν κάποια αξιοπρέπεια στην εξωτερική πολιτική, εσείς να ε, δεχτείτε ότι την καταστρέψατε. Στην συνάντηση της Γενέβης, εκεί θα είμαστε κομπάρσοι και σίγουρα όχι πρωταγωνιστές. Και τέλος απευθύνομαι σε εσά κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρόκ και σας ρωτάω, μήπως έχει έρθει η στιγμή στο πλαίσιο ευελιξίας της Επιτροπής μας να προβλέψουμε μια ειδική συνεδρίαση για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εγώ πιστεύω ότι έχει φτάσει πια η στιγμή να ανοίξουμε επίσημα ένα σοβαρό διάλογο τόσο για την εξωτερική πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για την εξωτερική πολιτική από πλευρά Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ, δεν θα αναφέρω τις, ε, δεν θα παραλάβω τα λόγια ανησυχίας των συναδέλφων, αλλά και για τις υπόλοιπες κρίσης, η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δεν ήταν δικαιολογημένη. Ούτε ανεκτή. Εδώ μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Τι ε, παράπλευρε συνέπειε θα υπάρξουν. Βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει, αλλά το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να ε, προκύψει ήδη αρχίζει να εξελίσσεται στο Λίβανο. Και στα κράτη του κόλπου και στην Τουρκία είναι υψηλό ο κίνδυνο και είναι σοβαρέ οι απειλέ. Τι προβλέπετε για την ευρύτερη περιοχή, γιατί είπατε ότι αυτό δεν συζητήθηκε ούτε τι θα γίνει με την Χεσμολά αν θα καταγραφεί στον κατάλογο τρομοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία. Εδώ ε, ε, λήφθη μια απόφαση για την αποστολή αρκετά προηγμένων όπλων στην Συρία και αυτό μα ανησυχεί ιδιαίτερω. Και τρίτε χώρε έχουν δεσμεύσει κάποιου πόρου για τη Συρία, αλλά δεν έχουν μεταφέρει τα χρήματα, όπω είπατε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ε, προβλήματα διαδικαστικά ε, για να λυθούν και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ανθρωπιστική κρίση. Θα εκτιμούσα λοιπόν να έχω τη σοφή σας τοποθέτηση σε αυτά τα θέματα. Κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Η πρώτη αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε όσον αφορά τους όρους μιας διεθνούς δυνατότητας να ασκήσει πίεση σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης τι γίνεται και πώς εκτιμάτε την κατάσταση σε σχέση με την έλλειψη απόφαση σε σχέση με την Συρία. Πώς υποβαθμίζει τη διεθνή μας κατάσταση, αν την υποβαθμίζει. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το εμπόριο όπλων. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν εργαλεία ή μέσα για να προλάβουμε το, να πάρουν ε, όπλα του καθεστώτος Ασάντ. Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ είμαι Λοιπόν, έχετε τον λόγο. I think it is important. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα το ότι η απόφαση που έπρεπε να ληφθεί και λήφθη την Δευτέρα ήταν μια απόφαση για την ανανέωση των κυρώσεων και της ανανέωσης του εμπάργου όπλων στη Συρία. Αυτή ήταν η απόφαση που έπρεπε να ληφθεί. Και όπως είπα δεν υπήρχε ομοφωνία να ανανεωθεί το εμπάργο όπλων στη Συρία στο σύνολό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η μορφή και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική από το Συμβούλιο με βάση τη συνθήκη και με βάση τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη να κάνουμε κάτι ή να μην μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Και όλοι μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας προσωπικά και τις έχουμε αυτές. Αλλά για το αν θα υπάρξει εμπάργο όπλων ή όχι, ή αν θα συνεχιστεί συνολικά το εμπάργο όπλων στη Συρία, ή αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή οτιδήποτε, Εκτός αν υπάρξει ομοφωνία, αυτή η απόφαση δεν μπορεί και δεν μπόρεσε να ληφθεί. Και δεύτερο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε, πώς να το πω, να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε στη σπουδαιότητά του και τη θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο τελικά. Να υποστηριχθεί δηλαδή η διαδικασία διαβουλεύσεων Γενέβης 2 και να εργαστούμε και συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα στεφθεί με επιτυχία η Σύνοδος Γενέβης 2 και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που πρέπει να είναι παρόντα να είναι παρόντα και να μην είναι κάποιο θαύμα μιας μέρας μόνο αυτό, αλλά να είναι μια αυθεντική διαδικασία, διεργασία που θα καταλήξει στο τέλος σε μια πολιτική ρύθμιση και συμφωνία και στην αποκατάσταση της ειρήνης για τους πολίτες, ε, τους κατοίκους της Συρίας. Και τρίτον, έχουμε και την κατάσταση όπου αντιμετωπίζουμε, πώς να το πω, το θέμα των προσφύγων, την ανθρωπιστική πλευρά του δράματος αυτού από πλευρά ΣΑΚ αναφέρθηκε το θέμα των επιπτώσεων στις γειτονικές ισόμορες περιοχές. Ναι, συζητήθηκε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί. Ο αριθμός των προσφύγων στην Τουρκία π.χ., στον Λίβανο, στην Ιορδανία πάλι εκεί. Και πολύ δύσκολες, δυσχερέστατες καταστάσεις που, υπό τις οποίες ζουν και διαβιώνουν οι πρόσφυγες εκεί. Εγώ είχα την ευκαιρία ο ίδιος να δω από πρώτο χέρι τους όρους και προϋποθέσεις διαβίωσης των προσφύγων στην Τουρκία. Σε μια κατάσταση που διαχειρίζονται καλά οι Τούρκοι, αλλά μια κατάσταση με μεγάλη ένταση για ευνόητους λόγους. Και επίση είχα την ευκαιρία από πρώτο χέρι τη Δευτέρα το πρωί να έχω μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Ένα θέμα δηλαδή με τον ε, Υπουργό ε, ε, των Εξωτερικών ε, Νταβούτογλου της ε, Τουρκίας. Ε, συζητήθηκε λοιπόν ε, το θέμα αυτό. Είναι γεγονός. Και το θέμα εξάλλου το οποίο αναφέρθηκε για το αν υπάρχει κάποιος τρόπος ίσως για τα όσα συμβαίνουν οι χώρες οι οποίες εξετάζουν να δώσουν όπλα στο καθεστώς Ασάν. Όχι, δεν υπάρχουν κάποιες τέτοιες χώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα από τα 27 κράτη-μέλη νομίζω σωστό είναι να πει κανείς ότι 25 δεν έχουν κανένα, καμιά πρόθεση να δώσουν όπλα σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους στη σύραξη στη Συρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα επιτόπου. Εκείνα τα κράτη που έχουν και θέλουν και εξετάζουν το να δώσουν όπλα θα πρέπει να το κάνουν υπό τους όρους και προϋποθέσεις ε, συγκεκριμένου καθεστώτος. Και αυτό το καθεστώς τι είναι, ποιο είναι. Πρώτον, συμμόρφωση Ευθυγράμμιση με τις θέσεις, τη θέση του Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων για την ΕΕ. Είναι η θέση του 2008. Δεν έχει μια άλλη κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι εξαγωγές όπλων να είναι ελεύθερη, ε, ελεύθερο εμπόριο για όλους. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τις εξαγωγές όπλων για την ΕΕ. Θεσπίστηκαν και ισχύουν από το 2008. Και αυτές οι αρχές, αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί εξακολουθούν και εφαρμόζονται και έχουν ισχύ. Και στη δήλωση που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ όλα τα κράτη-μέλη, όλα συμφώνησαν να συμμορφωθούν, να ευθυγραμμιστούν με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Οποιοςδήποτε θα ήθελε να επανέλθει σε σχέση με τις λεπτομέρειες αυτών των συμπερασμάτων θα δει ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα και ότι υπάρχουν αυτές οι αυστηρές αρχές, συγκεκριμένες αρχές και όροι για την ε, παροχή, για την ε, διάθεση όπλων στην ε, Συρία και μάλιστα με περιοριστικό χαρακτήρα, σε περιοριστικό πλαίσιο και επιπρόσθετα η διάθεση όπλων στη Συρία αποκλειστικά και μόνο αφορά την δέσμευση κρατών που θα επιθυμούσαν να το κάνουν. Αποκλειστικά και μόνο για τον συνασπισμό δυνάμεων της Συριακής Αντιπολίτευσης. Αποκλειστικά για την προστασία των πολιτών, των αμάχων και αποκλειστικά υπό και διασφαλίσεις που θα διέπουν αυτό το καθεστώς ε, διάθεσης όπλων. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα, ε, ε, όσα θα ακολουθήσουν. Γιατί οι πιο δυστυχή στη Συρία είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς ε, πρέπει να βοηθηθούν, που ζουν, διαβιώνουν υπό φρικαλές ε, συνθήκες και θα πρέπει να προχωρήσουμε και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας τώρα στο να μπορέσουν οι διαβουλεύσεις της Γενέβης 2 να ξεκινήσουν και να μεταξελιχθούν, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θετικό τρόπο. Όλοι να μπορέσουν να καθίσουν γύρω από την στρογγυλή τράπεζα εκεί στη Γενέβη 2 και να είναι μια, ε, ε, ένα γεγονός, ε, μια πρωτοβουλία, όχι μόνο διάρκεια μια ημέρα και τέρμα, αλλά να ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία θα στεφθεί στο τέλος με επιτυχία, με μια διευθέτηση για την εξέβρεση λύσης για την κατάσταση στη Συρία. Αυτό πρέπει να, πρέπει να τύχουν και αυτό πρέπει να κάνουμε οι πολίτες της Συρίας. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στόχος. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον Γενικό Γραμματέα, θα έλεγα. σα ευχαριστούμε εσά Γεια σα. Äh, θα ήθελα ε, να επαναλάβω ένα ερώτημα προς το Γενικό Γραμματέα. Τελικά, πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση της εξαγωγής όπλων. Ε, δηλαδή, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό να δημιουργήσει προηγούμενο, έτσι ώστε να εξαιρούνται τέτοιου τους πράξεις από την επιβολή κυρώσεων. Έχετε εσείς ε, κάποια άποψη από πλευράς υπηρεσίας εξωτερικής δράσης μετά από όλα αυτά που διαδραματίστηκαν. Πάρα πολύ σύντομα ε, θα ήθελα να προσθέσω ε, σε αυτά που μόλις τώρα είπε ο υπουργό ότι κατανοώ πολύ καλά τα αισθήματά σας και δεν είσαστε οι μόνοι και πολλοί άλλοι στο Συμβούλιο είχαν ε, την ίδια εντύπωση. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα πρέπει να το εξετάσουμε κάτω από τη σωστή σκοπιά. Ε, πράγματι ήρθε το εμπάργο όπλων και η απόφαση λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο όσον αφορά την κρίση στη Συρία. Δηλαδή ε, δεν ε, ισχύει αυτό για όλες τις αποφάσεις για το εμπάργο όπλων που λήθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Ο Υπουργό υπενήχθη την κοινή θέση του 2008, τον κοινό κώδικα Συμπεριφοράς και αν διαβάσετε αυτόν τον κώδικα θα εντυπωσιαστείτε από τα κριτήρια που περιλαμβάνει και που έχουν σχέση με όλο αυτό το θέμα της εξαγωγής όπλων. Βεβαίω στην περίπτωση της Συρίας, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, λόγω του ότι το εμπάργο όπλων ήρθε και επανήλθε η απόφαση στα κράτη-μέλη, εναπόκειται πλέον στους εθνικούς κώδικες να κρίνουν εκείνοι κατά πόσον ε, γίνεται σεβαστός ο ευρωπαϊκός ε, κώδικας ή όχι. Όμως τελικά τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν στο εγγύς μέλλον ότι ε, θα αποφασίσουν από κοινού για εμπάργο όπλων. Αν συμφωνήσουν και 27 και αύριο ας πούμε θα μπορούσε να υπάρξει επιβολή εμπάργο όπλων σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν ελήφθη απόφαση τη Δευτέρα επί της αρχής που να λέει ότι από τώρα και εφεξής οτιδήποτε έχει σχέση με εμπάργο όπλων είναι εκτός αρμοδιότητας της ΚΕΠΑ. Δεν ελέγχθη κάτι τέτοιο. Ε, η απόφαση αφορά μόνο, αποκλειστικά και μόνο τη Συρία. Βεβαίως η πολιτική δήλωση είναι σημαντική. Ακόμα και αν αποφασίζεται να επιτραπεί στην περίπτωση της Συρίας το ε, εμπάργκο όπλων να επανέλθει ως απόφαση τα κράτη-μέλη, αυτό έγινε, αλλά με βασικές, σημαντικές ε, ρήτρες ασφαλείας, όπως σας είπα, δηλαδή να γίνεται σεβαστός ο κώδικας συμπεριφοράς, επίσης ότι τα όπλα θα χορηγούνται μόνο ε, στον συνασπισμό επιτόπου για να προστατεύεται ο άμοχος πληθυσμός και επίσης και εγγυήσει ε, για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες αυτών των όπλων. Και κάτι άλλο, όπως είδατε στην πολιτική δήλωση, όλα τα κράτη-μέλη Ισραηλοί δήλωσαν ότι στη φάση αυτή δεν προτίθενται να στείλουν όπλα. Και τέλος θα υπάρξει και μία ρήτρα αναθεώρησης ε, σύμφωνα με την οποία οι Υπουργοί θα επανέλθουν στο θέμα αυτό πριν από το τέλος Ιουλίου. Γιατί τότε, γιατί ε, μέχρι τότε θα έχει φανεί πώς θα εξελίσσεται η διαδικασία της ε, Γενέβης. Αν δηλαδή τελικά ε, προχωρήσει καλά και σωστά η διαδικασία της ε, Γενέβης, τότε ενδέχεται να ληφθούν και άλλες ε, αποφάσεις από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και αν συμφωνήσουμε όλοι μας ότι δεν γράφτηκε πράγματι η καλύτερη σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό μας νομοποιεί αυτόματα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε άλλου είδους συμπεράσματα, γιατί η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαντάζεστε. Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω αυτό που διάβασα εχθές, μία ε, παρατήρηση ενός ε, πολύ καλού ιστορικού αναλυτή που έγραφε ότι αυτό που κατάφεραν την ε, Δευτέρα οι Ευρωπαίοι ήταν να αναγνωρίσουν ότι δεν συμφωνούν αλλά παρόλα αυτά μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό έγραψε. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν πριν ε, προβαίνει κανείς σε και κρίσεις για το τι έγινε τελικά τη Δευτέρα, καλό είναι να σκεφτεί κανείς ποια άλλη εναλλακτική λύση είχε μετά από 12 ώρες συζητήσεων όπου διαπιστώσαμε ότι ήμασταν διχασμένοι και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε επί της ουσίας ε, του θέματος. Η μόνη άλλη εναλλακτική λύση ήταν να ε, ακυρωθούν όλες οι κυρώσεις και θα βρισκόμασταν μπροστά σε μια κατάσταση με κανένα είδου κύρωση έναντι της Συρίας, πράγμα που θα ήταν πολύ χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν λάβαμε αυτή τη μεσοβέζικη απόφαση, επιτρέψτε μου να πω, που επιτρέπει όμως μια μετακίνηση. Και πρόεδρε θα πω και το εξή: αν δούμε λιγάκι τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν, αν τα διαβάσει κανείς ε, προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι εκεί ε, αναφέρονται πολλές ε, κατευθυντήριες γραμμές και διάφορα θέματα που διερωτηθήκατε κι εσείς όπως ας πούμε μεταπίδηση της κρίσης στο Λίβανο ή το θέμα των προσφύγων, της προσωρινής προστασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό και πολλά άλλα. Σε όλα αυτά τα θέματα προχωράμε και θα προχωρήσουμε περαιτέρω οι διπλωματικές μας προσπάθειες προχωρούν. Θα είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, με τη Ρωσία, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με διάφορους εταίρους μας και όλα αυτά θα προχωρήσουν μέχρι τη συνάντηση της Γενέβης. Και ελπίζω αυτή τελικά να αποδειχθεί μια ε, χρήσιμη διαδικασία. Η κυρία Γκόμες. Σημείωσα και έλαβα υπόψη προσεκτικά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα. Πρέπει, πιστεύω, να δούμε. Έχουμε μια έκθεση που βρίσκεται στην ΑΦΕΤ και πρόκειται να περάσει στην Ολομέλεια στη συνέχεια από ό,τι γνωρίζω για την υλοποίηση του Διοντολογικού κώδικα εξαγωγών όπλων. Νομίζω υπό το φως αυτής της, αυτών, αυτού του διχασμού και Τη διαίρεση στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να επανεξετάσουμε το περιεχόμενο αυτή της έκθεσης. Πρέπει εμεί νομίζω ω Ευρωκοινοβούλιο να στείλουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Ίσως υπάρχει η θετική αυτή ευμενής ερμηνεία που ο πρέσβης Λουμό μα έδωσε, αλλά μπορεί επίσης να υπάρχει και μια πιο αρνητική ερμηνεία ή θέση σε σχέση με μια οπισθοδρόμηση από αυτή τη συνέπεια για την κοινή μας θέση για τις εξαγωγές όπλων. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσεις στην ίδια τη Συρία, αλλά ίσως και πιο σοβαρές ακόμα επιπτώσεις πίσω και πέρα από τη Συρία. Γι' αυτό είναι ένας λόγος που πρέπει να μας κάνει να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα ως Ευρωκοινοβούλιο, αυτή την έκθεση ιδιαίτερα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το θέμα αυτό για την ομάδα επαφής. Δεν, δεν με ικανοποίησε η απάντηση που δόθηκε. Μια υπόθεση, ένα θέμα είναι η ομάδα δράσης για τη Γενέβη και το θέμα της Γενέβης και ένα άλλο θέμα είναι μια ομάδα επαφών των Ηνωμένων Εθνών όπου εκεί υπάρχει συν ε, υπευθυνότητα ε, για αυτά τα θέματα. Δηλαδή περί πρόκειται να κάνουμε τους Ρώσους και τους Κινέζους, την Ρωσία και την Κίνα για την λήψη αυτών των αποφάσεων το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών για την υπευθυνότητα, την ευθύνη να προστατέψουμε τους αμάχους στη Συρία να εμπλακούν και να είναι υπεύθυνοι να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν γίνεται αυτό σε σχέση με τη Συρία. Πρέπει να έχουμε συναγάγει τα συμπεράσματα από προηγούμενες κρίσεις και να μπορέσουμε να δράσουμε σωστά. Και σε σχέση με την αναφορά στον ε, πρέσβη ε, Λαχντάρ Μπραήμι δεν μπορεί να αυτό να επαρκεί και σε σχέση με την ομάδα επαφών να δούμε αν μπορεί κάτι να ενισχύσει, να ενδυναμώσει αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν το κάναμε αυτό. Τέλος, Λιβύη συνδέεται με το θέμα της ε, σφαιρικής ολοκληρωμένης προσέγγισης για το θέμα του Μάλι. Το γνωρίζουμε αυτό. Αναγνωρίζοντας όμως ότι μέχρι σήμερα δεν είμαστε και ιδιαίτερα τρομερά επιτυχείς θα υπάρχει και υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέλλον γι' αυτό, διότι έχω πλέον κουραστεί με αυτούς τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών που πάνε και έρχονται ασταμάτητα. Ε, σε ευχαριστούμε κυρία Άννα Γκόμες. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και πάντα πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός και γνωρίζω φυσικά ότι πολλοί ε, αισθάνονται στο Συμβούλιο όπως και εμείς σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργό Εξωτερικών τη Αυστρία βγήκε έξω και είπε στον γερμανόφωνο τύπο ότι πρόκειται για μια αποτυχία, δεν συμφωνήσαμε. Μετά ξαναπήγε στην αίθουσα και συνέχισε τις διαπραγματεύσεις. Ήταν λοιπόν, ας το πω έτσι και στο επαγγελματικό επίπεδο του Συμβουλίου, ολέθρια η κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε και το θέμα της λειτουργικότητας των ε, διαδικασιών στο Συμβούλιο που δεν είναι και ε, το καλύτερο. Όμως έχοντας ακούσει αυτά που είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ιρλανδία ότι κανένα δεν μίλησε για εθνικό συμφέρον, δύσκολο είναι να το πιστέψω αυτό, γιατί αυτό έκανε ο Βίλιαμ Hague. Μίλησε για εθνικά συμφέροντα σε σχέση με το, ε, το εθνικό ακροατήριο. Τώρα, αυτό είναι όμως το θέμα και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω εδώ είναι αυτή η δήλωση. Είναι μια δήλωση όπου διακηρύσουμε και λέμε ότι θα συμμορφωθούμε και θα ευθυγραμμιστούμε με τον νόμο. Ουσιαστικά η Γαλλία και η Βρετανία τι συμφώνησαν να μην λέει παραβούν τον νόμο. Εξαιρετικό, ε, συγχαρητήρια, υπέροχο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μας κάνει να αγνοήσουμε ότι αυτό ήταν ένα σοβαρότατο λάθος. Και τελευταίο, το οποίο θα πρέπει και αυτό να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, είναι να περάσουμε σε μια πιο σοβαρή θεμελιώδη συζήτηση. 12 ώρες για μια τέτοια συζήτηση είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και στο τέλος αυτής της συνάντησης Έχω πάει, έχω παρακολουθήσει τέτοιες συνεδριάσεις. Υπάρχει μόνο η επιλογή μεταξύ δύο κακών, αρνητικών επιλογών. Αλλά δεν μιλάμε και δεν κάνουμε λόγο για αυτές τις 12 ώρες. Κάνουμε λόγο για δύο χρόνια, διετή περίοδο. Με τη Λιβύη ήταν ανίκανη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει από κοινού. Η Βρετανία και η Γαλλία κινήθηκαν ως πρωτοπόροι. Μαλή, κάτι έπρεπε να γίνει εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ικανή να δράσει. Η, η Γαλλία ε, κινήθηκε ως προπομπός, ως πρωτοπόρος. Στη Συρία δεν υπάρχει συμφωνία. Πάλι δύο κράτη είναι εκείνα τα οποία υιοθετούν μια θέση και έχουμε μια ξεχωριστή κατάσταση. Λοιπόν, η ευρύτερη πρόπτικη με κάνει και ανησυχώ ιδιαίτερα για την ΚΕΠΑ για το μέλλον και την προθυμία των κρατών μελών μας με σοβαρό τρόπο να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή πορείας και πλεύσης όταν έχουμε κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμό για τις επεξηγήσεις που μας έδωσε. Νομίζω ότι έθεσε σαφώς το πρόβλημα. Το σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και πιστεύω ότι οι επεξηγήσει του είναι σκόπιμες και επικοδομητικέ. Και ούτε πρέπει να κάνουμε το λάθο να είμαστε μαζοχιστέ, αναζητώντα ενόχου στο Συμβούλιο Υπουργών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα εκεί που τίθεται με όλη την ομότητα και σκληρότητά του και την προβληματική που συνεπάγεται είναι στο Συμβούλιο ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών προφανώ όπου υπάρχουν μέλη, δύο μέλη με δικαίωμα αγνησικηρίας που δεν υλοποιούν τι υποχρεώσει του. Και τρίτο στοιχείο Νομίζω ότι ακολουθούμε τελείω λάθος πορεία στη συζήτηση αν αυτό το εξηγήσουμε και το θεωρήσουμε μια κατάσταση που θα μα κάνει να εξετάζουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων των κρατών μελών για την ομοφωνία ή όχι. Αυτό που αναζήτησε το Συμβούλιο είναι αναζήτησε λύσεις σε ένα σοβαρό προφανές πρόβλημα όπου καθημερινά όπω είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ιρλανδία, υπάρχουν θύματα άνθρωποι που δολοφονούνται και υπάρχουν πρόσφυγες και φυσικά πόσοι είναι εκείνοι που πεθαίνουν και σκοτώνονται ενώ εμείς συζητούμε Πιστεύω ότι το να μην συζητήσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε λόγο για διεκδικήσεις και απαιτήσει των κρατών μελών και να επιβάλλονται θέσεις ε, κρατών μελών στο σύνολο των υπολείπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια λανθασμένη ερμηνεία. Οι πολίτες αναμένουν από εμά και αναμένουν από το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης να είμαστε σε θέση να βρούμε λύσεις στα προβλήματα. Και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να δράσουμε. Εκεί ακριβώς πρέπει να κάνουμε κάτι για την ε, επίμαχη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανατίθεται στα κράτη-μέλη το να αποφασίσουν τι θα γίνει με το θέμα των κυρώσεων όσον αφορά το εμπάργο όπλων. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο το οποίο είναι η θέση του, μέσα στο πλαίσιο των κανόνων και ρυθμίσεων που έχουμε θεσπίσει. Αλλά δεν πρέπει να καταλήξουμε σε μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων και να ξεχάσουμε τα πραγματικά προβλήματα στα αναμένουν οι πολίτες να δοθούν λύσεις, να σταματήσει δηλαδή η σφαγή των αμάχων στη Συρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά καλωσορίζω τα λογικά σχόλια, εχέφρανα σχόλια του κυρίου Ντομό. Και για να απαντήσω στον κόμιτα, στον κόμι Λάμστορφ για την επίθεση κατά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί δεν ευθυγραμμίστηκα σε σχέση με την ΚΕΠΑ. Δεν θυμάμαι να έγινε κάτι τέτοιο για τη Γερμανία σε σχέση με τη μη ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις για τη Λιβύη από τη Γερμανία. Και η πραγματικότητα είναι, όχι μόνο σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η πραγματικότητα είναι δεν υπάρχει κάτι σαν μία ενιαία και μόνη ΚΕΠΑ. Υπάρχει μία ΚΕΠΑ την οποία συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη, επί τη οποία συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη. Πάντα υπό τι αρχέ των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και η Γαλλία και η Βρετανία θεώρησαν ότι η λιγότερο επώδυνη λύση θα ήταν να εξοπλιστούν ε, οι αντιπολιτευόμενοι ε, των Ασάντα να μπορέσουν να αποκτήσουν όπλα. Ε, ελπίζοντα ότι θα υπάρξει ένα είδο ε, κάποτε μια ε, φεντεραλιστικής πολιτικής ε, που πόρο απέχει. Εμείς ε, προκειμένου με την τάση που υπάρχει να εγκαταλείψει η Βρετανία την, Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε δράσεις της ΚΕΠΑ μέσα σε ένα ευθετό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ έχω μια πρόσθετη ερώτηση. Ίσως το συμπέρασμα το τελικό μπορεί να είναι λαθασμένο από πλευρά μου. Η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία τι κάνουν θα το είχαν ρισκάρει οι οικονομικές κυρώσεις να μπορούσαν να είχαν ε, αρθεί όσον αφορά αν, αν δεν είχαν γίνει αρκετά σε σχέση με τις ε, εξαγωγές όπλων. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα ποια θα ήταν η κατάσταση ή ποια θα ήταν, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα σε σχέση με τις διαβουλεύσεις. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι όλοι θα είχαν, θα ρισκάρει όλες οι άλλες κυρώσεις να είχαν αρθεί και να είχαν οδηγηθεί σε μια διαφορετική κατάσταση. Πρόεδρε, αν μπορείτε να με αφήσετε να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις σύντομα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτός ακριβώς ήταν ο κίνδυνος. Αν εκείνοι που δεν ήθελαν να προχωρήσουν στο να άρουν το εμπάργο όπλων αποφάσιζαν ότι δεν υπήρχε πλέον συμφωνία και εγκατέλειπαν την αίθουσα. Δεν θα υπήρχαν πλέον κυρώσει ή εμπάργο όπλων. Γι' αυτό την 11η ώρα και πράγματι την 11η ώρα των διαβουλεύσεων είναι αυτό που μας έκανε να αποφασίσουμε ότι θα έπρεπε να βρούμε κάτι το οποίο θα ήταν μια ήπια προσγείωση, μια δυνατότητα προσγείωσης ήπιας, μια δυνατότητα δηλαδή να, μπορέσουν, να μπορέσουμε να δούμε αν θα μπορούσαν να αρθούν ε, οι ε, κυρώσεις σε σχέση με τους αμάχους και να αφήσουμε στο ε, πλάι το εμπάργο όπλων. Αλλά αυτό θα απαιτούσε ομοφωνία. Θα έπρεπε πάλι να υπάρξει ομοφωνία για να εγκριθεί κάτι τέτοιο. Γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτό. Τόσο απλό ήταν το θέμα επ' αυτού. Τώρα, απαντώντα στην παρέμβαση τη Αναγκόμες για τη Γενέβη, αυτό πίστευε είναι το πρόβλημα το οποίο είδαμε ότι ε, έπρεπε να μπορέσει να γίνει. Ήταν μια διάσκεψη η Γενέβη, όχι μόνο διάσκεψη, αλλά και ομάδα επαφής για τη δράση μας. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς μας υποστηρίζαμε την διεργασία της Γενέβης κατά της βούλησης όλων των ε, υπόλοιπων εταίρων στη διεθνή κοινότητα. Πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Αυτό που ξεκίνησε στην ε, Γενέβη το, στις 30 Ιουνίου 2012 δεν ήταν ένα συμβιβασμός για να υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση στη Συρία. Ήταν η προσπάθεια να μπορέσουν τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, οι πέντε του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, και επτά άλλες χώρες, Ιράκ, Τουρκία, Κατάρ και κάποιε άλλε χώρες συν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση αυτού του συμβιβασμού. Ποτέ δεν καταφέραμε να ε, συγκαλέσουμε πάλι αυτή την ομάδα γιατί κάποια μέλη αρνήθηκαν να προσέλθουν. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Στι 30 Ιουνίου εκείνοι οι οποίοι ήταν παρόντε σε αυτή τη συνάντηση δεν ήταν πλέον πρόθυμοι να το ε, ξανακάνουν και να δώσουν συνέχεια σε αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό πήρε ένα ολόκληρο χρόνο και αυτό με οδηγεί στην παρέμβαση του κυρίου Σαλαφράγκα. Ένα χρόνο και 80.000 νεκρούς κόστησε για να αποφασίσουμε στο τέλος τέλος ότι η Γενέβη ήταν το εύθετο πλαίσιο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Αν δεν κατανοήσει κάποιος αυτό το σκηνικό, αυτή την προϊστορία, δεν θα μπορέσει να κατανοήσει το πώς ε, οδηγηθήκαμε στο να κατακαιρματιστούν τα κράτη-μέλη. Διότι δεν ήταν η ορθή ε, πορεία να υπάρξει συνέχεια χωρίς να ε, δοθεί συνέχεια στη Γενέβη. Πρέπει λοιπόν να ξαναξεκινήσει η διεργασία Γενέβης και πρέπει να, ξε... να προωθηθεί. Και υπήρξε συμφωνία ότι ελπίζω ότι θα την υλοποιήσουν και θα τηρηθεί για να ξαναξεκινήσει αυτή η διεργασία της ε, Γενέβης. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τώρα ένα τελευταίο στοιχείο να προσθέσω για αυτό που είπε ο κύριος Λάμστοφ για τη Λιβύη, το Μάλι και τη Συρία. Κατανοούσε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λάμστοφ και νομίζω ότι αληθεύει ότι όταν συζητήσαμε τα θέματα, συζητώντα τα θέματα και πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη. Αλλά εδώ να κρούσω κόδωνα κινδύνου, να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι τρει αυτέ κρίσει διαφέρουν τα μέγιστα, τα μάλα η μία από την άλλη. Στο Μάλι, όπω σωστά αναφέρατε, είμαστε σχετικά καλά προετοιμασμένοι στο να υπάρξει κάποια δράση ε, από πλευράς ε, ε, πρωτοπόρου δράσης ε, με την διπλωματική δράση το νέο ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη για μια ομάδα ειρηνοποιών και από πλευρά της Αφρικής κιόλας ε, ειρηνοποιού ομάδας. Έτσι προχώρησε η διεργασία. Αυτό που άλλαξε ήταν το ότι όλοι εξεπλάγησαν με την απόφαση των επαναστατών να ξαναπάρουν τα όπλα και να κινηθούν κατά της κυβέρνησης στο Νότο και να κινηθούν κατά του Μπαμάκο. Ίσως θα έπρεπε να το είχαμε προβλέψει αυτό. Ίσως οι υπηρεσίες ε, κατασκοπία σε πληροφοριών θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει και να το έχουμε λάβει αυτό σε σχέση με την προετοιμασία ε, της δράσης μας. Μπορεί να είναι σωστό να το πείτε αυτό, αλλά το να πει κανείς ότι δεν έγινε τίποτα και ότι υπήρξε μια άρνηση από τα κράτη-μέλη να εξεταστούν δυνατότητες δραστηριοποίησης μέσα στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ δεν είναι ο σωστός τρόπος να το θέσει κανείς αυτό. Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε αυτό. Με τη Λιβύη όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη. <clears throat> Κάποιοι συμμετείχαν, κάποιοι όχι από τα κράτη-μέλη. Αλλά με τη Συρία ας δούμε την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να λάβει μια απόφαση όσον αφορά τη στρατιωτική συνιστόσα. Είναι το σύνολο της διεθνούς κοινότητας που έχει αμφιβολίες και προβλήματα για το πρακτέο, για το τι πρέπει να γίνει και διστάζει η διεθνής κοινότητα και πρέπει να συζητήσουμε και τα θέματα της επιβολής μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, τα θέματα ανθρωπιστικής ε, διάστασης και όλα αυτά στη συζήτηση και στη ΣΥΠΑ και στα Ηνωμένα Έθνη κάθε φορά το θέμα ήταν ε, προβληματικό για την λήψη απόφασης. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση να διεξαχθεί και να ληφθούν αποφάσεις. Πολύ περίπλοκα και σύνθετα τα προβλήματα. Και βλέποντας και τις αποφάσεις της Δευτέρας, δύο ερμηνείες, δύο αναγνώσεις μπορούν να υπάρξουν επ' αυτών, που πάλι καταδεικνύουν και πρέπει να δείχνουν ότι συζητώντα τα θέματα της Συρίας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για την αξιολόγηση και τις ε, ε, αποφάσεις, οι ερμηνείε. Ε, που λαμβάνονται. Είναι μια πολύ ρευστό κατάσταση. Αλλάζουν τα πράγματα άρδιν από τη μία στιγμή στην άλλη σε σχέση με μια κατάσταση και μια άλλη. Μακρηγόρησα πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενικέ Γραμματέα για το ότι παραμείνατε μισή ώρα περισσότερο και μπορέσαμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ε, και σίγουρα δεν την ολοκληρώσαμε. Σας εύχομαι τα καλύτερα και σας ευχαριστώ πολύ.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 Κυρία Αντρικίνε, έχετε να κάνετε παρατηρήσεις επί της έκθεσης. Ε, όχι κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να κάνω καμία παρατηρήση. Μπορούμε να ε, προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία αμέπως αμέργο, όπως λέμε. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Πρόεδρε, ε, κύριε Λάμπστροφ, αυτό λέει πρώτος είναι δικό σας πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Ε, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έκλεισε. 33-6 εγκρίθηκε η τροπολογία. Η απόφαση της κυρίας Λάμστοφ δεν παίζει κανένα ρόλο κύριε Λάμστοφ. Λοιπόν πάμε στην επόμενη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 ήταν αυτή. 23 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία, στην συμβαστική 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 50 υπέρ κατά ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά ή μάλλον σηκώστε χέρι 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 52 και η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ή 57. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 60. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61. Υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 73 μισό λεπτό, έχει καταπέσει 73, πάμε στην 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 12 υπέρ Τροπολογία 12 παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η ψήφο σας, ε, κύριε Λάμψοφ, και πάλι δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν είναι καθοριστική. Η 14 υπέρ Μισό λεπτό. Η 13 πρώτα. Η 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 14 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Κύριε Λαμπστόφ, ε, η ψήφο σα πάλι και δεν παίζει κανένα ρόλο. Απορρίπτεται έτσι κι αλλιώ. Συμβαστική 3 παρακαλώ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογίε 1 και 2 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνονται, η 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική επαλήθευση έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπέρ, τα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Die Abstimmung ist geschlossen. Έκλεισε η ψηφοφορία. Κύριε Λάμπστο, τι είστε υπέρ ή κατά. Υπέρ εγκρίνεται λοιπόν με δύο εποχές. Έτσι λοιπόν εγκρίνεται η έκθεση. Σας συγχαίρουμε κυρία εισηγήτρια. Η ε, ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Και πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Λαμπστόφ για τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, ποιος θα αναλάβει την ε, Προεδρία, ο Στάνθος κύριος Προβέρμπα. Προβέρα. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Κύριε Λάμπστοφ, έχετε το λόγο. Jetzt, jetzt auf einmal habe ich das Wort. Τώρα δηλαδή μου δίνετε το λόγο. Αυτό. ευχαριστώ. Γίνεται κάποια φασαρία στην αίθουσα. Να περιμένω λίγο μέχρι ότου οι συνάδελφοι συγχάσουν Να τελειώσουν τις συζητήσεις τους. Για τον λόγο κύριε ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα, να επεξηγήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάσσεται αυτή η έκθεση. Πρόκειται για μια σύσταση προ το Συμβούλιο για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα ξεκινήσει όπω και τα προηγούμενα έτη. Πρόκειται για μια εργασία που με μεγάλη συνένεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων προχωρεί και υλοποιείται. Ησυχία παρακαλώ. Έχουμε εδώ και κάποια χρόνια μια θεσμοθετημένη μορφή διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για αυτά τα θέματα. Και επίσης εδώ και κάποια χρόνια τακτικά πάει μια αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ βρισκόμαστε σε μια διεργασία που ετήσια επαναλαμβάνεται. Ωστόσο όμως με διαφορετικά κέντρα βάρους ε, εκπεριτροπής εκάστοτε. Και σήμερα με αυτό το ψήφισμα ή το σχέδιο σύστασης έχουμε για παράδειγμα και το θέμα τοποθέτησης σε σχέση με τη συμφωνία με το Διεθνές Εμπόριο Όπλων σε σχέση με τα όσα είχαν τα Ηνωμένα Έθνη αναλάβει ως πρωτοβουλία. Είναι ένα επίκαιρο θέμα που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Για μας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ποιο ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε και τη συζήτηση για τη στάση των δύο αυτών μελών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια περίπλοκη εικόνα Τώρα, η έκθεση αυτή θεωρεί και εξετάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, παγκόσμιο, παγκόσμια, σκηνή εμπλεκόμενο για ε, αυτά τα θέματα έχει δίκιο ο συνάδελφο Παντσέρη σε σχέση με αυτά. Πρέπει επί των αρχών να εξετάσουμε το τι συμβαίνει. Περνάμε στο τμήμα ειρήνη και ασφάλειας ε, για την ανάπτυξη μέσα σε πλαίσια δράσης, δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, σε πεδία δραστηριοποίηση. Είχαμε χθε μια συνάντηση όπου από τις 108 τροπολογίες που κατατέθηκαν καταλήγουμε, καταλήξαμε σε κάποιες νέες συμβιβαστικές τροπολογίες που εκπονήθηκαν και εδώ ακολουθήθηκε η διεργασία ότι από κοινού συνεργαστήκαμε ώστε να μπορέσουν έτσι να διαμορφωθούν οι συμβαστικές τροπολογίες ώστε να είναι αποδεκτές από τις πολιτικές ομάδες. Εκφράζω την ικανοποίησή, μου για το ότι τα καταφέραμε. Μία τροπολογία συζητήσαμε εξειδικευμένα που κάπως τροποποιήσαμε εναντί της περσινής χρονιάς. Είναι το θέμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, την υποστήριξη του εκδημοκρατισμού με την αποστολή αποστολών και ομάδων παρατηρητών εκλογών. Είχαμε και έχουμε την κατάσταση ότι ενοχλούν δεν πολλές φορές οι ειρηνοποιοί και δεν γνωρίζουν τι θα γίνεται και τι μπορεί να γίνει επί τόπου με μια τέτοια αποστολή παρατήρησης εκλογών και πώς θα διαμορφώνονται αυτά τα πλαίσια. Είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο εμβαθύνουμε μέσα στο πλαίσιο της ομάδας Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου και εκλογές με κάπως τροποποιημένο τρόπο φέτος έναντι της περσινής χρονιάς. Βρήκαμε όμως καλή διατύπωση για όλα αυτά. Όλα αυτά με μια κοινή προφορική ερώτηση θα διαμορφωθούν και ελπίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί αυτή η προφορική ερώτηση. Όσον αφορά τον πίνακα ψηφοφορία για αύριο, προσπάθησα όλα αυτά θεματολογικά με ένα ενιαίο πλαίσιο, σε ένα ενωμένο πλαίσιο να τα διατηρήσουμε. Υπάρχουν σημαντικά θέματα που μπορούν να συζητηθούν. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν σε σχέση με τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, σύμβαση για εμπόριο όπλων, το θέμα των offsets να ε, εξεταστεί, να συνενταχθεί. Ένα, είναι ένα οικονομικό πολιτικό θέμα και όχι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο το, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία που έχουμε παραδοσιακά από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα μακροσκελές τμήμα για τις διεργασίες αυτές σε σχέση με την ε, νέα μεταξέλιξη των στόχων της χιλιετίας της, ε, ε, για την ανάπτυξη και την αηφορία. Η Επιτροπή Ανάπτυξη σίγουρα θα συντάξει μια ξεχωριστή έκθεση από πλευράς της που θα συμπεριλαμβάνει αυτά τα σημεία ώστε να μπορέσουμε αυτή την ε, πτυχή τον ε, Νοέμβριο να την έχουμε ολοκληρώσει και με τους εταίρους μας να την προαγάγουμε. Έχουμε κάτι το καινούριο θεσμικά σε αυτή τη διεργασία και έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την πτυχή. Και αυτό είναι το αίτημα προς το Συμβούλιο εμείς μετά τη Γενική Συνέλευση να ξανασυνέλθουμε και να ξαναδούμε ποιες προτεραιότητες είναι αυτές ε, που εντοπίσαμε και ταυτοποιήσαμε, με ποιο τρόπο ε, υπήρξαν επιτυχίες και τι συνέβη με την ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ή που δεν υπήρξαν οι ε, αυτές, αυτές ε, δράσεις που να στέφθηκαν με επιτυχία. Ένας κύκλος δηλαδή που πρέπει να ολοκληρωθεί σε σχέση με αυτά τα θέματα που τον διάλογο μεταξύ του Συμβουλίου της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δώσει την δυνατότητα μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με αποτελεσματικό τρόπο να καλύψουμε αυτά τα θέματα. Χαίρομαι σε σχέση με τη συζήτηση αυτών των θεμάτων ε, με την ομάδα εργασίας για τα θέματα των Ηνωμένων Εθνών μετά τις ερνές διακοπές που να τα ξανασυζητήσουμε. Προσβλέπω στα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας τώρα. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κόμι Λάμστορ για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους σκιώδεις εισηγητές και εξίσου να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με τους συμβιβασμούς, τις συμβαστικές τροπολογίες που αποφασίσαμε, εγκρίναμε χθες. Νομίζω οι συμβαστικές τροπολογίες βελτιώνουν και με σαφή τρόπο βελτιώνουν τις συστάσεις μας προς το Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Υπογραμμίζουν, τονίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Φυσικά Ιδιαίτερα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με μια ενιαία ενωμένη φωνή να τοποθετείται σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει και γενικό πλαίσιο σύστασης για τα θεσμικά θέματα, αλλά και αναφορά στα επίκαιρα θέματα, όπως την Συρία ή το Μάλι όπου φυσικά η διεθνής κοινότητα πρέπει να μπορεί να παρέμβει και να αναλάβει δράση. Το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε χθε έχει επεκταθεί, έχει διευρυνθεί με αρκετά άλλα θέματα, ακόμα και την συμφωνία για το εμπόριο όπλων, για παράδειγμα, ως σημείο αναφορά. Πρέπει επίσης να προσθέσω κάτι εδώ και να πω ότι τα κράτη-μέλη μέσα στο πλαίσιο αυτών την 1η Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να κυρώσουν αυτή την συμφωνία. Δυστυχώς την τροπολογία 74 της κυρίας Γκόμες δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Η κυρία Γκόμες τι ζητεί. Ζητεί πέρα από το πλαίσιο αυτής της ε, συμφωνίας ε, να μπορέσει να αναλυφθεί δράση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Εξίσου εκφράζω την λήψη μου για το γεγονός ότι ο εισηγητής στην δική μου τροπολογία υπαριθμών 26 δεν την υποστηρίζει. Διότι πιστεύω εδώ συγκεκριμένα ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε αρκετά παραδείγματα που καταδείκνυαν ότι αν δεν υπάρχει συνένεση, συμφωνία με ομοφωνία τουλάχιστον εκείνα τα κράτη που πλειοψηφικά υιοθετούν κάποια θέση πρέπει να μπορούν να, να την υλοποιήσουν. Θα μου άρεσε, θα με ικανοποιούσε αν οι τροπολογίες 1137, 93 και 98 μπορούσαν να, να εγκριθούν. Ωστόσο, επίσης έχω και μια τροπολογία ενός συναδέφου, την τροπολογία 88 δηλαδή εδώ, που αναφέρεται στον αντισημιτισμό. Θα μπορούσε να είχε παραμείνει στο κείμενο, να είχε ενταχθεί σε αυτό. Κατά τα άλλα όμως το σχέδιο έκθεσης είναι ισορροπημένο, είναι ισόρροπο και Θεωρώ ότι η ψηφοφορία αύριο θα μπορέσει να καταδείξει ότι συμβαίνει αυτό και ότι θα το δεχτεί και θα το προαγάγει. Ευχαριστώ. Για παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και για τις προσπάθειες του κυρίου Λάμστορφ ε, για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο από πλευράς Ευρωβουλής ε, για τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και κάποια προληπτική, ας το πω έτσι, απογοητευτική τοποθέτηση σε σχέση με μια χήμερα, το να υπάρξει δηλαδή ε, να παρουσιαστεί μια θέση ενιαία και μια ενιαία τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό στις Βρυξέλλες, πώς μπορεί να γίνει στη Νέα Υόρκη. Και σε σχέση με τα θέματα της ε, των συμβαστικών τροπολογιών συμπεριλαμβάνουν την πλειοψηφία των προτάσεών μας από της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας και όσον αφορά και τις επιφυλάξεις ε, που έχουν εκφραστεί για την συνεκτικότητα και την συνολική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη να αναζητηθεί και να προασπιστεί μια κοινή θέση των κρατών μελών στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ Ο εγκάρσιος χαρακτήρας της ε, συνιστώσας του φίλου σε όλες τις διαδικασίες πρόληψης και επίλυσης σειράξεων είναι ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε σχέση και με τη σύραξη στη Συρία παρόλη την πραγματικότητα ως έχει, ζητούμε να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε ευθύνη και να προστατεύσουμε τους αμάχους στην ανθρωπιστική δράση, την οικονομική υποστήριξη των προσφύγων και σε σχέση με την κατάσταση της Σαχέλ και την κατάσταση στο Μάλι η πρόταση συμμετοχή ε, συμμετοχής στις ε, ε, δράσεις υπέρ της ειρήνης για την ειρηνοποίηση. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις, κάποιες διαφορετικές τοποθετήσεις όσον αφορά τη φιλελεύθερη ομάδα και το ΕΛΚ για τη σπουδαιότητα που έχει για μας τους σοσιαλιστές η σύμβαση για το εμπόριο όπλων και σε σχέση με την 74 της κυρίας Γκόμες. Το αίτημά μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει έναν μηχανισμό εποπτείας για την μεταφορά όπλων την καταπολέμηση του θολού χαρακτήρα της αδιαφάνειας στο εμπόριο όπλων και μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως ε, είναι κάποιοι ίσως εναντίον μιας μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την εξαγωγή όπλων. Όταν έχουμε υπό ενδυνάμει μια, ε, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας σύμβασης ε, για την εξαγωγή όπλων και σε σχέση με τις τροπολογίες 86 και 96 του Ραϊμόνο Μπιόλς που αναφέρονται στην αναγνώριση στην αναγνώριση σε σχέση με την βία που ασκείται κατά των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων, των εκπροσώπων, των ομοφιλοφίλων και των λεσβιών. Ε, εδώ το θέμα πρέπει να είναι και σε σχέση και με αυτά τα θέματα στην παράγραφο 1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είχαμε μια λιγική θέση και μια πιο συναφή και συνεκτική θέση με την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην τροπολογία 92 ζητείτε να δοθεί κύρια προτεραιότητα στην κατάργηση της θανατικής ποινή παγκόσμια. Και δεν ξέρουμε γιατί έχουν αρνητικό πρόσημο στον πίνακα ψηφοφορία σας και οι δύο τροπολογίες. Ιδιαίτερα σε σχέση και με την τροπολογία 91 όταν έχουμε ε, ε, τη διαφορά μεταξύ τους. Και ολοκληρώνω Πέρυσι εγκρίθηκε στη σύσταση η ανάγκη να υπάρξει η ισορροπία μεταξύ της ομάδας των 20 και της δράσης σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και σε σχέση με την έλλειψη προόδου προς, αυτό, αυτή την κατεύθυνση μας εκπλήσει ότι εφέτος ο εισηγητής είναι εναντίον. Και επίσης εγκρίναμε τον όρο των κλιματικών προσφύγων, προσφύγων λόγω των κλιματολογικών αλλαγών. Και σε σχέση με τους ε, στόχους που πρέπει να είναι δεσμευτικοί όσον αφορά την πολιτική μας ε, μέχρι το 2020 και θέλουμε να δειχθεί υποστήριξη στις τροπολογίες της ομάδας μας σε σχέση με τα κύρια αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών. Μία ε, δράση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς του 2003 που υπεγράφει και κυρώθηκε από τα κράτη-μέλη και, όλα τα, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, για τη χώρα μου έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλά να πω ότι από ό,τι φαίνεται ε, εμείς έχουμε διαφορετική απαριθμίση των τροπολογιών. Είπατε 96 για τους ε, ομοφιλόφιλους. Για μας όμως είναι το περιβάλλον. Μπερδεύτηκαν κάπως οι τροπολογίες και 86 δεν έχουμε εμείς μπροστά μας οι σοσιαλδημοκράτες την ε, ίδια ρύθμιση τροπολογιών, ε, γιατί αναφέρονται κάποια θέματα που νομίζω ότι είναι λίγα και επίμαχα. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Βότσον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μου κύριο Λαμπστόφ για τη δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Νομίζω είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που έχουμε κάποιον ο οποίος παρακολουθεί με τέτοιο ζήλο τις σχέσεις ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω στους συναδέλφους ε, ε, μια τροπολογία που έχω καταθέσει με διακομματική υποστήριξη. Νομίζω ότι μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας σχετικά με τη σύσταση κοινοβουλευτικής συνέλευσης για τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η τροπολογία στη διατύπωσή της είναι πολύ προσεκτικοί, θέλουμε να προσελκύσουμε την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Δεν προτείνεται άμεση αλλαγή, αλλά τουλάχιστον προτείνεται να ε, προβληθεί αυτή η ιδέα του να υπάρξει κοινοβουλευτική συνέλευση στο πλαίσιο μεταρρύθμισης ενός οργανισμού, ο οποίος ε, άντεξε θαυμάσια ε, στο διπλωματικό τομέα, προσέφερε πολλές υπηρεσίες και έχει υποφέρει από εθνικές προσεγγίσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όσοι βρισκόμαστε εδώ, συνάδελφοι όπως ο κύριος Πέτερινγκ, ο οποίος ε, παρακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως άμεσα εκλεγόμενο σώμα. Όλοι μας λοιπόν γνωρίζουμε τη συμβολή του Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση προς την εξέλιξή του μιας πολιτικής οντότητας. Ε, τα κοινοβούλια διαφέρουν από οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο συνενώνουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται όχι μόνο να εκπροσωπούν συμφέροντα της γενέτηράς τους, αλλά και να προάγουν κοινά συμφέροντα στο φορέα που βρίσκονται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, έχουμε την ε, διακομματική υποστήριξη για αυτή την τροπολογία. Δεν περιμένω οικουμενική υποστήριξη. Ε, ξέρω ας πούμε ότι ο κύριος Τάνοκ ή άλλοι θα φρίξουν με την ιδέα ότι θέλουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική συνέλευση για τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά τουλάχιστον ελπίζουμε να έχουμε την υποστήριξη των, περαιτέρω, των περισσότερων με σε αυτή μας την ε, τροπολογία. Ο κύριος Τάνοκ, ε, κοιτάξτε, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύετε για μένα, εγώ στηρίζω αυτή την αρχή που προβάλλατε. Και μάλιστα το είχα δείξει κιόλας, αλλά δεν ήσασταν παρόν ε, στην αρχή της εβδομάδας ε, που ήρθε εδώ εκπρόσωπος των ΟΜΕ και είπε ότι καταρχήν ε, το θέμα είναι οικονομικό. Ποιο θα πληρώσει, γιατί θα είναι ακριβό το να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι βουλευτές να πηγαίνουν στη Νέα Υόρκη και να γυρίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το δεύτερο είναι ότι περίπου το 50% των ε, κρατών ε, μελών των ΗΠΑ δεν είναι κοινοβουλευτικέ δημοκρατίες. Τώρα πιανού κοινοβούλιο θα αναγνωρίσετε και πιανού όχι. Ποια χώρα ναι και ποια χώρα όχι. Επίσης, ναι, είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, για τη μερικοί που θα έρθουν αυτοί θα ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να υπερασπιστούν τα προσωπικά τους ε, συμφέροντα. Ας πούμε, από την Καμπότζη. Αλλά και πάλι εγώ ε, πιστεύω στη δημοκρατία, πιστεύω στα κοινοβούλια και όσο και αν σας φαίνεται οξύμορο, εγώ στηρίζω την πρότασή σας. Να πω απλώς ότι σε αυτό το πλαίσιο ο πατριωτισμός μου, και παρακαλώ να το σημειώσετε αυτό, ο πατριωτισμός και όχι εθνικισμός μεταβάλλεται σε μία απόλυτη αφοσίωση το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τη μόνιμη θέση του στη Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Αθνών και μάλιστα να είναι μια αγία προτεραιότητα αυτή, καθαγιασμένη από παρά όλα όσα λέγονται από συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή ε, και στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως, οι εργατικοί συνάδελφοι κατά την προεκλογική εκστρατεία λένε ότι θα τα αφήσουμε αυτά με την ε, μόνιμη θέση ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου στο ε, ΝΟΙΕ. Πολύ ξεκάθαρη απάντηση και τώρα να απαντήσει ο εισηγητή. Δεν θα αμφισβητούσε σε καμία περίπτωση τον πατριωτισμό του Λόρδου Ντάρτμουθ Απλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ των ομάδων σε σχέση με όσα λέει η έκθεση, ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε την μόνιμη δεσμευσή μας και ότι θέλουμε και μια μόνιμη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Είναι ενδιαφέρον που χρησιμοποιήθηκε ο όρος ε, καθαγιασμένο μιας από τις παλιότερες ε, δημοκρατίες στο πρόσωπο της γης με θρησκευτικές και πολιτικές ελευθερίες. Αλλά είναι το αγαπημένο μας σημείο που μας αρέσει να διαφωνούμε. Δεν μπορούμε παρά να ακολουθήσουμε την άποψη της πλειοψηφίας εδώ και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει στήριξη για την συνολική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει με μεγάλη ταχύτητα σε τέτοιες μέρες, σε τέτοιους καιρούς διότι υπάρχει ενθουσιασμό στην ομάδα των πέντε για μεταρρύθμιση, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μαριάν, να συμφωνήσω, θα πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα, διότι ορισμένα θα πρέπει να τα δούμε και πάλι με λεπτομέρειες, για να ελέγξουμε και την αρρύθμιση, τη σωστή αρρύθμιση των τροπολογιών. Ίσως μπερδεύτηκα εγώ, ίσως δεν άκουσα καλά για την κοινοβουλευτική συνέλευση. Η συζήτηση αυτή επαναλαμβάνεται κάθε φορά, κάθε χρόνο. Είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε με μεγάλη προσοχή και διεξοδικά για το τι πρακτικές ε, συνέπειες μπορεί να έχει. Και επίσης ε, πόσο μπορεί να επηρεάσει ενοιολογικά. Υπάρχουν κάτι μέλη που συμμετέχουν στα Ηνωμένα Έθνη και υπάρχει και σχετική χάρτα που καθορίζει τη συμμετοχή των και των μελών στη Γενική Συνέλευση. Τίποτε, απολύτως τίποτε στην χάρτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να στέλνουν βουλευτές στις εθνικές αντιπροσωπίες. Πολλοί κάνουν ε, ακριβώς αυτό. Όταν πηγαίνει υπουργό εξωτερικών και ε, οι συμμετέχοντες ε, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν ταυτόχρονα και στην Γενική Συνέλευση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε ένα σώμα που ενώνει βουλευτές και συνδυάζει τα δικά τους συμφέροντα και προτεραιότητες με αυτά των Ηνωμένων Εθνών. Πολλοί έχουν καθεστώς παρατηρητών. Νομίζω λοιπόν ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση απλώ θα επαναλάβει τα όσα κάνει η Γενική Συνέλευση και κάτι άλλο που έχει πάλι σχέση με τη Χάρτα. Εάν μια Κοινοβουλευτική Συνέλευση δημιουργηθεί <clears throat> βάσει τη Χάρτα, θα πρέπει να έχει καθεστώ παρατηρητή, έστω και από μακρού, ή θα είναι ένα επικουρικό ε, όργανο, υποβοηθητικό της Γενικής Συνέλευσης. Άρα οι βουλευτές, ως προς το νομικό τους ε, καθεστώς, θα έχουν μειωμένο κύρο σε σχέση με τους διπλωμάτες που εκπροσωπούν ε, τις κυβερνήσεις και τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Γενική Συνέλευση. Καλό είναι μπορείτε να σταθμίσετε αυτά μέχρι να αποφασίσουμε και να δούμε πώς θα ψηφίσουμε σχετικά. Για τους πόρους, σχολιάστηκε και αυτό. Είναι ένα ζήτημα που παραδοσιακώς δεν το έχουμε επιλύσει, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός καταμελών μελών των ΗΠΑ που πραγματικά δεν είναι, είναι κάθε άλλο παρά δημοκρατικά. Θα βρούμε ως Ευρωκοινοβούλιο τους εαυτού μας, θα τους φέρουμε σε πολύ δύσκολη θέση διότι υπό την οπτική γωνιά του, ΟΗΕ είμαστε ένα σώμα περιφερειακής ολοκλήρωσης όχι κάποιου κράτου. Αλλά τι θα γίνει με του δημοκρατικά εκλεγμένου Βορειοκορεάτε συναδέλφου ή με του Κινέζου συναδέλφου, του δημοκρατικά εκλεγμένου Κουβανού συναδέλφου, οι οποίοι θα ισχυρίζονται ότι ω βουλευτέ μπορούν να καθορίσουν την πορεία των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό ω σήμερα δεν έχω πιστεί ακόμη ότι είναι εύστοχο να έχουμε κοινοβουλευτική συνέλευση. Είναι πολύ συνετό διατυπωμένη η τροπολογία σα. Δεν είναι συντηρητικά διατυπωμένη, βρίσκω κύριε Βότσον, γιατί δεν είναι ταυτόσιμε αυτέ οι έννοιε. Αλλά γιατί να θέλουμε τόσο πολύ μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Εγώ θα βάλω ένα μείον στον κατάλογο ψηφοφοριών, όπω είχα κάνει και τα περασμένα έτη. Βεβαίω ο κάθε συνάδελφο μπορεί να αποφασίσει μόνο του τι θέλει να ψηφίσει, αλλά νομίζω ότι να ενδυναμωθεί η Γενική Συνέλευση και να βελτιωθεί η συνεργασία των συναδέλφων στο επίπεδο τη ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι το καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουν τα Ηνωμένα Έθνη σωστά. Περιμένω λοιπόν την ψηφοφορία αύριο και να ανυπομονώ να συνεργαστώ με του συναδέλφου στα πλαίσια τη ομάδα εργασία για το θέμα. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Επόμενο σημείο. Θα πρέπει να κλείσουμε μέχρι τι 11.30, σωστά. Διότι θα έρθει ο Πρωθυπουργό τη Σερβία. Θα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό τη Σερβία. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομοι από τώρα από τον κύριο Γκάλερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ε, ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών στο Πακιστάν στις 14, 7-14 Μαΐου 2013. Στις 11 Μαΐου οργανώθηκαν εκλογές και ήταν ιστορικό γεγονός, γιατί ήταν η πρώτη φορά που από το 1947 μια κυβέρνηση ελεύθερων πολιτών ε, μετέφερε την εξουσία σε μια άλλη ελεύθερη κυβέρνηση. Οι εκλογές θεωρήθηκαν σχετικά ε, ελεύθερες και δίκαιες με ποσοστό συμμετοχής 60% το υψηλότερο από το 1970 ε, και να δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για να μας ενημερώσει σχετικά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα κάποιου αριθμού και κάποια γεγονότα να αναφέρω. Και στην αξιολόγηση θα μιλήσω αγγλικά στη συνέχεια, διότι τα στοιχεία είναι όλα διαθέσιμα στα αγγλικά για αυτά. Η αποστολή στις 3 Απριλίου με την ε, ομάδα μας κατέληξε στο Ισλάμ, στο, στο και στις 4 Ιουνίου θα κλείσει τις ε, πύλες και στις 2 Ιουλίου, την εβδομάδα της Δευτέρας Ιουλίου, θα έχουμε την τελική έκθεση με συστάσεις δικές μου που θα μπορέσουν να παρουσιαστούν σχετικά. 52 μακράς διάρκειας παρατηρητές σε 26 ομάδες είχαμε και 46 σύντομης ε, διάρκειας παρατηρητές ε, είχαμε με τους διπλωμάτες επιτόπου και μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου είχαμε πάει σε ε, πολλά τμήματα υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ ε, Χάουιτ ε, και είχαμε και δύο άλλους συναδέλφους. Κάποια λίγα στοιχεία δεν χρειάζεται σε σχέση με να έχει κανείς φόβο. Δεν συμβαίνει τίποτα με τους μακράς διάρκειας παρατηρητές. Τα τελευταία στοιχεία που είναι διαθέσιμα τι λένε. Δείχνουν ότι συνολικά 46,2 εκατομμύρια εκλογής ε, κατέληξαν στα εκλογικά κέντρα και 55% δεν ήταν 60% 55% συμμετοχή στις εκλογές ε, αυτές έναντι 44% τις προηγούμενες εκλογές ε. Είναι λοιπόν ε, αυτά κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι είναι μια σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε. Διαφορετική η συμμετοχή στις εκλογές στην πρωτεύουσα Ισλάμαμπατ 62%, 60% στη μεγαλύτερη επαρχία στο Παντζάμπ, στο ε, Σίντ στη συνέχεια και στο Κάιμπερ Παστούν 45% ε, στο Βελουχιστάν Κέτα πρωτεύουσα 43% πρωτεύουσα του Μπελουτσιστάν και στις ομοσπονδιακά διαχειριζόμενες ε, περιοχές και φιλετικές περιοχές 36% συμμετοχή στις εκλογές. Δυστυχώς την ημέρα των εκλογών ε, κάποια βία σημειώθηκε που οδήγησε σε ε, νεκρούς 64 θύματα σε σχέση με την εκλογή ε, ε, οι βιοπραγίες αυτές. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε και σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες γίνεται ακόμα καταμέτρηση, υπάρχει, πρέπει να γίνουν επανεκλογές σε κάποιες περιφέρειες εκεί όπου κέρδισαν σε άλλες περιφέρειες και έπρεπε σε περίπτωση απόφασης να είναι υποψήφιοι και σε άλλη εκλογική περιφέρεια να γίνουν επανεκλογές. Δεν έχουν αποφασιστεί ε, οι εκλεγμένοι σε όλες τις περιφέρειες. Το PMLN του Ναουάζ Σαρίφ είναι ο μεγάλος νικητής ε, που ε, έχουν τις 72 ε, έδρες από τις άμεσες εκλογές 140 ε, συνολικά κέρδισαν η μεγάλη χαμένη είναι το Λαϊκό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν Pakistan People's Party με 31 έδρες από 0 σε 28 έδρες κατέληξε ο Ιμραν Χάν ο παίκτη του κρίκετ με το PGI με 28 έδρες το Περιφερειακό Κόμμα στο Καράτσι που παραδοσιακά είναι ισχυρό στο Καράτσι 18 έδρες ε, κέρδισε και ένα Ισλαμικό κόμμα Τζαμάτ JUIF ε, είναι η σύνμηση απέξε 10 έδρες όλα τα άλλα κόμματα κατέληξαν σε κάτω από 10 έδρες είναι αξιοπρόσεκτο ότι το Awami National Party συνολικά μόνο μία έδρα κατάφερε να αποκομίσει από αυτές τις εκλογές για τη χρονική διεξαγωγή. Μέχρι τις 26 Ιουνίου θα έχουμε τις, τη διαδικασία των επανεκλογών. Μάλλον πρόκειται για 7 έδρες στην Εθνική Συνέλευση. Η συγκρότηση σύνοδος θα είναι την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τις 3 Ιουνίου, μέσα σε αυτές τις 3 μέρες δηλαδή, θέλουν να εκλέξουν και τον Πρωθυπουργό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο Ναουάζ Σαρίφ ο νέος πρωθυπουργός του Πακιστάν. Και τώρα περνάω στα αγγλικά διότι έχουμε τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που θα ήθελα να παρουσιάσω και δεν θα ήθελα να παρεκκλίνω από τις διατυπώσεις που έχουμε στα κείμενά μας στα αγγλικά. Αξιολογήσαμε και θεωρήσαμε ότι η εκλογική διαργασία ήταν ε, αποδεκτή παρόλες τις ε, ε, βιοπραγίες και τις κάποιες ελλείψεις που υπήρξαν. Κάποια από τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν ότι θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε μια σημαντική δέσμευση για τον εκδημοκρατισμό από τα κόμματα και που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ότι έχει διαπιστωθεί ε, σε διάφορα μέρη της χώρας, δηλαδή στο Καράτσι, την ίδια την πόλη και στο Μπελουτσιστάν, στο Κάιμπερ Παστούν και όπου σημειώθηκαν κάποιες ε, πράξεις βίας ε, και σε σχέση με την συμμετοχή στις εκλογές ήταν υψηλότερη στο Παντζάμπ από ό,τι αλλού. Είχαμε ένα συγκεκριμένο σημείο ότι οι Ταλιμπάν του Πακιστάν καταρχήν είχαν δηλώσει ότι οι εκλογές δεν είναι Ισλαμικές και δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν οι πολίτες σε αυτές με τη συμμετοχή από 44% σε 55% των πολιτών στην εκλογή καθοριστικά μπορούμε να πούμε τελεσίδικα δεν υποστήριξαν αυτή την προσέγγιση των Ταλιμπάν οι πολίτες του Πακιστάν και επιπλέον είχαμε μια στοχοθετημένη ή συγκεκριμένη απειλή κατά τριών κομμάτων που θεωρήθηκαν κόμματα κοσμικού χαρακτήρα το εθνικό το Ασβάμι και το NPM στο Καράτσι. Εναντίον τους οι Ταλιμπάν είχαν δηλώσει και το έκαναν και στην πράξη στο θέτησαν κάποιους υποψηφίους και συναντήσεις αυτών των κομμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα κόμματα απόλεσαν τον ένα ή άλλο υποψήφιο και στη συμμετοχή σε συναντήσεις ή συνεδριάσεις. Δεν μπόρεσαν πλήρως δηλαδή να ολοκληρώσουν τις προεκλογικές συναντήσεις τους στο μέτρο όπως το είχαν προσχεδιάσει. Η δημοκρατική πρόοδος του Πακιστάν μπορεί να εξεταστεί στην ε, αύξηση όσον αφορά τις εκλογές με περισσότερα κόμματα που συμμετείχαν και πάνω από διπλάσιους υποψηφίους όσον αφορά τις εκλογικές περιφέρειες. Η παρατηρητές ε, των εκλογών ε, σε μεγάλα τμήματα της χώρας ε, όπου παρακολούθησαν τις εκλογές σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κόμματα τα οποία είχαν ζητήσει να υπάρξει κάποιο μποϊκοτάζ και σε σχέση με τον Μπελουτσιστάν, τους εθνικιστές του Παστούν, αυτή τη φορά συμμετείχαν στις εκλογές. Και το θέμα πρέπει να ε, εξεταστεί σε σχέση με την απειλή των εθνικιστών διότι είναι ε, εκείνοι που θέλουν να αποσχιστούν από το Πακιστάν και είχαν οδηγηθεί σε κάποιες ε, βίες πράξεις διότι δεν ήθελαν να, να ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο. Ένας ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αύξηση των υποψηφίων γυναικών. Υπερδιπλασιάστηκαν. Επίσης υπήρξε και ένα σύστημα για την ε, σχέση με τον διαχωρισμό των ε, ψήφων όσον αφορά ε, γυναίκες και άνδρες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά εκλογικά κέντρα στο Πακιστάν για άνδρες και γυναίκες είτε τελείως ξεχωριστά αναφύλλω, είτε σε σχέση με ένα εκλογικό κέντρο ξεχωριστές, ξεχωριστή ψήφιση για άνδρες, ξεχωριστή για γυναίκες και βλέπουμε ότι σε σχέση με τις υποψηφίους ε, και σε σχέση με το χαμηλότερο ποσοστό παρόλη την προσπάθεια που έγινε 86 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ε, καταχωρηθεί. 11 εκατομμύρια είναι λιγότερες οι γυναίκες από ότι οι άνδρες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί για την δυσαναλογία αυτή. Για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, οι γυναίκες έχουν 60 πρόσθετες θέσεις ε, που δεν ε, ε, εκλέγονται άμεσα αλλά μέσω της ε, αναλογικής αυτής εκπροσώπησης και με τον καθορισμό των εδρών αυτών για τις έδρες αυτές με τα αποτελέσματα σε σχέση με τα κόμματα αναλογικά οι έδρες όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών κατανέμονται στα κόμματα ανάλογα δηλαδή με τις θέσεις που ως απόθεμα πρέπει να εκπροσωπούν γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για την εκπροσώπηση των μη μουσουλμάνων με τις ε, θέσεις που καταχωρούνται για αυτούς. Τώρα, σε σχέση με την τελευταία φορά, τι συνέβη κύρωσε το Πακιστάν την ε, ε, σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτές είναι οι πρώτες εκλογές ε, που διεξάγονται υπό τις υποχρεώσεις που έχει πλέον το Πακιστάν για αυτό το θέμα. Και εμείς με την εφαρμογή αυτών των κανόνων ως, εκλογή, ως αποστολή παρατηρητών, δηλαδή υπάρχουν οι απαιτήσει για να είναι κάποιο υποψήφιο. είδαμε μια εξέλιξη που δεν ήταν τόσο σημαντική την τελευταία φορά που είχαμε πάει εκεί το 2008 για τις εκλογές. Δύο ε, κανονισμοί σε σχέση με το Σύνταγμα, τα άρθρα 62 και 63 όσον αφορά την ε, ε, εκπροσώπηση από πλευράς υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια και τα πιο υποκειμενικά είναι για παράδειγμα αν, αν είναι κάποιος καλός μουσουλμάνος ή όχι και αυτό με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίστηκε από εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για την καταχώρηση των υποψηφίων όσον αφορά τις διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Έπρεπε να εξεταστεί αν είχαν όλοι δικαίωμα να είναι υποψήφοι σε αυτές τις εκλογές. Είδαμε κάποιες αξιοπερίεργες αποφάσεις που ελήφθησαν, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά πολλές φορές ανατράπηκαν κάποιες αποφάσεις για την εκπροσώπηση, για την υποβολή υποψηφιωτήτων από πλευράς αυτών των ατόμων. Επίσης ε, όσον αφορά μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την ε, ε, δυνατότητα των εκλογών εκπροσώπηση στο Πακιστάν, αυτοί οι μηχανισμοί αποτελεσματικά εφαρμόστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, παλαιότερα και την τελευταία φορά ο κύριος εκλογικός επίτροπος με διάταγμα διοριζόταν από τον πρόεδρο είχαμε μια αλλαγή και ήταν μια σύσταση από την τελευταία φορά να υπάρξει μια κοινοβουλευτική επιτροπή που θα καθορίσει τον επίτροπο αυτό και στο τέλος ομόφωνα θα αποφάσιζαν για τον ε, εκλογικό επίτροπο διακομματικά μέσω μιας συμφωνίας που θα λαμβανόταν από αυτούς. Είναι μια σημαντική πρόοδος που συνεισφέρει υπέρ της αξιοπιστίας υπέρ της αξιοπιστίας της εκλογικής ε, ε, διαδικασίας. Να μπορέσει δηλαδή η Επιτροπή αυτή διακομματικά, υπερκομματικά να δράσει. Ως προς αυτό το στόχο νομίζω ε, μπόρεσε να επιτευχθεί λόγω της συνενετικής αυτής διαδικασίας τον διορισμό του κύριου εκλογικού επιτρόπου για τις εκλογές. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. Ωστόσο ναι, σας ζητώ να ολοκληρώσετε λέει ο Πρόεδρος, να ολοκληρώσετε γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές, κάποια άλλα θέματα τα οποία βελτιώθηκαν παρότι όχι προ πλήρη ικανοποίησή μας ε, ο ρόλος των εκλογών ήταν ε, διαφανής αυτή τη φορά. Δεν υπήρξαν ισχυρισμοί ώστε να, έχουν, ε, να θεωρείται ότι υπήρξαν κάποιες παρατυπίες και επίσης ε, καταρχήν ε, οι δημοσιογράφοι είχαν περισσότερο πεδίο ελεύθερης δράσης, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι μπόρεσαν εξίσου να καλυφθούν όλα τα κόμματα. Γνωρίζουμε από στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ότι και στην δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε σχέση με το κόμμα της αντιπολίτευσης ε, που είχε τη μεγαλύτερη κάλυψη. Μετά ακολουθούσαν ο Ιμραν Χάν και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν, α το πούμε έτσι, ένα δίκαιο πεδίο δράσης όσον αφορά το, τα μέσα, της, ε, μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμως δεν οφείλεται σε κάποια παρέμβαση, επέμβαση από πλευρά της κυβέρνησης, αλλά σε διαφορετικές επιλογές όσον αφορά ε, τους ιδιοκτήτες των διαφορετικών τηλεοπτικών σταθμών για την κάλυψη των υποψηφίων. Η κοινότητα των Αχμάντι εξακολουθούσε να υφίσταται αρνητικές διακριτικές ε, ρυθμίσεις ε, σε σχέση με ένα ξεχωριστό ε, εκλογικό ρόλο που στο τέλος οδήγησε σε μποϊκότ όλων αυτής της κοινότητας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσε να καλυφθεί επαρκώς. Ολοκληρώνω εδώ και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή λεπτομέρειες θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Κύριος Χάουιτ παρακαλώ, εσείς. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ο μιλητής μιλάει χωρίς μικρόφωνο. everybody. Democracy is, of course. Η δημοκρατία ε, είναι καλά οργανωμένη στην Ευρώπη, γι' αυτό και συζητάμε ε, σήμερα για το Πακιστάν. Ε, για αστείο το είπα, ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ο μιλητή ο κύριος εισηγητής παλαιότερα και θα θυμάται από τότε ότι αυτά που είπε επηρέασαν τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, συναδέλφους ε, οι οποίοι ε, με συνόδευσαν στην αποστολή. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι πήγαμε στον Ουκαλάνη δέκα μέρες πριν από τις εκλογές και εκεί έγινε μία ομιλία με βάση την οποία ε, είχαν δηλώσει ότι δεν θα επέμβει ο στρατός και θα υπάρξουν δημοκρατικές εκλογές. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε ότι στη χώρα αυτή η δημοκρατία είναι εύτραυστη, όμως οι εκλογές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Όσον αφορά τη βία, είχαμε μία συζήτηση για το πώς ε, μπορούμε να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό. Η βία από μόνη της ε, βεβαίως και είναι φρικιαστική και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Ε, οι Ταλιμπάν στο Πακιστάν έχουν στοχεύσει σε τρία κόμματα ε, και αυτό ίσως επηρέασε το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Υπήρξε μια ε, δραματική συνάντηση με τους Ταλιμπάν. Οι άνθρωποι αυτοί ε, είχαν μαζί τους και τα όπλα. Ε, μερικοί αναφέρθηκαν σε επιθέσεις των Ταλιμπάνων που σκοτώθηκαν πάρα πολλοί πολιτικοί εκπρόσωποι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήταν μια ξεκάθαρη ψήφος ε, των Πακιστανών κατά αυτών των απειλών. Ανέφερε ο κύριος Γκάλερ τα σχετικά ε, στοιχεία στον Παλουτσιστάν. Εκεί έχουμε μια περιοχή όπου γίνονται πολλές επιθέσεις και όπου οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να εκφοβούνται. Ένα από τα πράγματα που επιθυμώ να προβάλλω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι αν διαβάζουμε μόνο τα ευρωπαϊκά μέσα για τη βία στη χώρα δεν αποκτούμε σωστή εικόνα της κατάστασης. Εγώ πήγα στο Πουντζάπ. Εσείς ε, μιλήσατε για αστείες εκλογές, ενθουσιώδεις εκλογές, ε, οι άνθρωποι συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό το παρατηρήσαμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η δέκατη φορά που παρατηρώ εκλογές και για πρώτη φορά ε, διαπίστωσα ότι υπήρχαν ε, υπόνοιες για ε, νοθεία. Σε τελική ανάλυση όμως ε, δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η υποψία. Στο Καράτσι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Το γεγονός όμως ότι υπήρχε επιτροπή παρατηρητών, αυτό ήταν ήδη από μόνο του ένα καλό σημάδι. Για μένα η δημοκρατία παγιώνεται καλύτερα αν δει κανείς το τοπικό επίπεδο της τοπικές εξελίξεις. Ε, οι άνθρωποι θέλουν να υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή ανάμεσα στους ε, ψηφοφόρους και τους ε, πολιτικούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουμε. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα πω δύο πράγματα. Όσον αφορά τις ευρύτερες επιπτώσεις αυτών των εκλογών είναι σαφές ότι η σταθερότητα στη χώρα είναι καθοριστική σημασία για όλους μας για λόγους ασφάλειας και διότι είναι μια μεγάλη χώρα με στρατηγικό εμπόριο, με επιρροή στην επιροχή και στην περιοχή και ευρύτερα. Εγώ νομίζω ότι ε, μοιάζει να προκύπτει σταθερότητα, μια σταθερή πλειοψηφία από τις εκλογές. Δεν έχω δει ποτέ ένα σύστημα που να μπορεί κανείς ε, με το κινητό του τηλέφωνο ε, να βρει ε, που είναι το εκλογικό του τμήμα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό ε, στον κόσμο. 14 εκατομμύρια χτυπήματα είχαμε με αυτό το σύστημα, μοναδικό το σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε όχι μόνο για το Πακιστάν αλλά και για άλλες χώρες. Και βεβαίως ε, κάτι το ιδιαίτερα δυσάρεστο όπου ε, τις τελευταίες μέρες εξαρτίας ένας από τους αρχηγούς ήταν στο νοσοκομείο υπήρξε όμως ε, μία συγκέντρωση πολλών οπαδών του και τα είδε μέσα από βίντεο link και αυτός συνδέθηκε με πλατφόρμα γιγαντοοτόνη για να ενθαρρύνει τους οπαδούς του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι οι εκλογές αυτές μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα, ε, βλέποντας όμως ε, τον ε, κώδικα συμπεριφοράς των εκλογέων, αυτό και μόνο αρκεί. Πάντως ε, θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους συναδέλφους να εκφράσουν την άποψή τους. Για μένα θεωρώ ότι ήταν τεράστιο προνόμιο να συμμετάσχω στην ε, Επιτροπή Παρακολούθησης Εκλογών στο Πακιστάν. Ε, το απόλαυσα και ήταν πολύ πιο θετικό από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Ευχαριστώ τον Μάικλ και όλους τους συναδέλφους που έδωσαν τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει τόσο σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια και προς τον κύριο Γκάλερ, ο οποίος δεύτερη φορά ανέλαβε τέτοια αρμοδιότητα και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Ήταν μεγάλο το θάρρος τους να αναλάβουν μια τέτοια αποστολή, διότι υπήρχαν απειλές, απειλές βίας από τους Ταλιμπάν και άλλους εξτρεμιστές που δεν πιστεύουν ε, καταρχήν στην ε, δημοκρατία και την εκλογή κυβέρνηση μέσω της κάλπης. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν σημαντική η, διασφάλεια, διασφάλιση της προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρώτη φορά λοιπόν δημοκρατική μετάβαση από μια κυβέρνηση σε μια επόμενη με συνθήκες ειρήνης, ασφαλείας και δημοκρατίας σημαντικότερες για όλη την περιοχή, την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη. Τώρα δεν ήθελα να θέσω ένα πολιτικότερο ερώτημα για την νέα κυβέρνηση του Πακιστάν, γιατί μας αφορά και εμάς. Έγινε ένα σχόλιο από τον νέο Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρίφ, ότι έμαθε από τα διδάγματά του όταν εκδιώχθηκε από τον Μουσάραφ ε, το στρατιωτικό καθεστώ της χώρας. Λέει ότι ήταν όριμος ω υποψήφιο. Και διερωτώ με, επειδή είμαι μεγάλο φίλο τη Ινδία και βρίσκω πολύ καλή αυτή την εξέλιξη. Έγιναν σοβαρέ δηλώσει για την επιθυμία του να εμβαθύνει, να προσεγγίσει έτσι περαιτέρω την Ινδία, να επιληθεί το θέμα του Κασμίρ και να δημιουργηθούν δύο βιβλία επικοινωνία ώστε να ξεπεραστεί η ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα αναφέρει ότι θέλει να αρχίσουν συνομιλίε με του ε, Ταλιμπάν του Πακιστάν. Του μετριοπαθέστερου δηλαδή Ταλιμπάν αυτό θα γίνει και στην πράξη. Ήταν κάτι που οργανώθηκε ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία. Και ποιες είναι αυτές οι συνιστώσεις των Ταλιμπάν που είναι περισσότερο ορθολογιστικές. Και τι θα γίνει και με τις ανάλογες περιοχές της Ινδίας. Και για τους χριστιανούς ε, ε, του Πακιστανούς στο Λονδίνο αλλά και τους Ινδουιστές και τις σχέσεις τους τι ε, σχέση υπάρχει με τις, μειονότη... με τις μειονότητες και πώς σκοπεύει να τις καλύψει με την κυβέρνησή του ο νέος ε, πρωθυπουργός, ο εισηγητής για τις απαντήσεις. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου θα ήθελα να κάνω και μια τελική παρατήρηση μετά την ε, τελική έκθεση και τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και πρόγραμμα παρακολούθησης για να συνεργαστεί ξανά και περισσότερο με τις νέες αρχές, το νέο κοινοβούλιο, τη νέα εφορευτική επιτροπή, για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Η συνεργασία λοιπόν αυτή τη τελευταία πενταετία πρέπει να εξακολουθήσει. Υπάρχει πολιτική βούληση και θα πρέπει να τη δώσουμε την κατάλληλη όθηση για να σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα. Ω προ τα υπόλοιπα σημεία μετά τι εκλογέ, και αφού κατέστη σαφές ότι ο κύριο Σαρίθα ήταν ο Πρωθυπουργό, προσεκάλεσε μέχρι και τον ε, ε, Ινδό για να παραστεί στην ανάληψη καθηκόντων. Στην ανάληψη καθηκόντων του. Ανέφερε και την ε, αναμενόμενη απόσταση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν Και βεβαίω ήταν πολύ πιο εύκολο να περάσουν από το Πακιστάν τα αμερικανικά στατεύματα από ότι αεροπορικό. Κοιτάξτε κύριε Γκάλερ, είναι εδώ ο Πρωθυπουργό. Μου είπατε δύο λεπτά. Τέλο πάντων. Νομίζω. Θα, δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Mr. Κύριε Χάουιτ. Μα Όσα είπε ο κύριο Τάνοκ για τι μειονότητε χριστιανών, ήταν σημαντικό ότι ο κύριο Σαρίφ πριν τι εκλογέ, σε συνέντευξη, σε ενδό δημοσιογράφο για την ειδική τηλεόραση, είπε ότι κάποιοι τον επικρίνουν εντό του κόμματό του, αλλά θεωρεί συμβολικό σημαντικό να προσεγγίσει την Ινδία. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και για του Ταλιμπάν του Πακιστάν, είναι μια σαφής απειλή και υπήρξαν και επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών. Υπάρχει όμως καταδίκη από την κοινή γνώμη και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Υπάρχει καλύτερος συσχετισμός μεταξύ Ταλιμπάν του Πακιστάν και του Αφγανιστάν αλλά η διεθνή κοινότητα ε, λέει πια ότι πρέπει να συζητήσουμε με τους Ταλιμπάν. Πρέπει να διαπραγματευτούμε μήπως και βρεθεί μια πολιτική λύση. Οι Πακιστανοί πολιτικοί με το ίδιο πνεύμα προσέγγισαν τα πράγματα. Κύριε Χάουιτ, σας παρακαλώ. No problem. Συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Yes, we receive the Prime Minister. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση με το σημείο υπερθμών 9 της ημερήσιας διάταξης. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω σήμερα εδώ από κοινού τον συνάδελφό μου Έντουαρτ Κούκαν, τον επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας, τον κύριο Ιβίτσε Αιντάτσιτσε, τον Πρωθυπουργό της ε, Δημοκρατίας της Σερβίας, από τον Ιανουάριο ε, βιώσαμε πάρα πολλές εξελίξεις. Η συμφωνία με το Κοσμοπέδιο είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και επίσης σημαντικό είναι και το πρόγραμμα εφαρμογής. Σας συγχαίρω για την προσωπική σας ε, αφοσίωση, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό έχει προκύψει κάποια δυναμική. Επίσης, χαίρομαι που επιθυμείτε να διασφαλιστεί η θέση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. με είδαμε τους τελευταίους μήνες να λαμβάνονται μέτρα κατά της ε, διαφθοράς. Σημαντικό αυτό όπως και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ο αγώνας κατά της ε, ε, διαφθοράς και της εγκληματικότητας είναι καθοριστικά στοιχεία και αποτελούν τη βάση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προσβλέπουμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ιουνίου. Είμαστε πεπισμένοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι τελικά θετικό θα προκύψει αίσιο τέλος. Ελπίζω λοιπόν ότι η θέση που έχετε ε, λάβει, τα επιτεύγματα που έχετε να επιδείξετε, όλα αυτά μας ε, οδηγούν στο σωστό δρόμο. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολλές ε, σημαντικές ιστορικές πλευρές του θέματος που αφορούν την ουσία του κράτους σας. Ε, ε, αν αυτά επιληθούν ηρωνικά, αυτό θα αποδείξει και το δρόμο που ακολουθείτε και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε ε, τις, τις, την παρέμβασή σας, την εισήγησή σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε Μπρόκ. Κυρίες και κύριοι, ε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για το ότι με προσκαλέσατε να κάνω αυτή την παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου ευθύ εξ αρχής να παρουσιάσω και να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το πρόσφατα εγκεκριμένο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο για την ένταξη ως προοπτική της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Σερβίας και νέα όθηση δίνεται στην κυβέρνησή μας να δώσουμε συνέχεια στην πορεία μας προς την Ευρώπη. Κατά το τελευταίο διάστημα έκανε σημαντικά βήματα η Σερβία στο να διασφαλίσει αυτό το ευρωπαϊκό της μέλλον. Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ε, ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, ελήφθησαν με ιδιαίτερη σοβαρότητα υπόψη για να δοθεί μια ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προ ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο για μα είναι ένα ρεαλιστικό και εφικτό στόχο. Κυρίε και κύριοι, Υιοθέτησε τον διάλογο με την Πρίστινα, με το Κωσυφοπαίδιο η Σερβία στο ανώτατο επίπεδο με τη διαμεσολάβηση της ΥΠΑ της εκπροσώπου αρμόδιας για την ασφάλεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίας Κάθη Άστον καλοπροαίρετα και με την βούληση να ε, προσεγγίσουμε μακροπρόθεσμα λύσεις προς το αμοιβαίο συμφέρον που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και με μεγάλο πολιτικό ρίσκο η Σερβία κατάφερε να υλοποιήσει, να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία με την Πρίστινα, διασφαλίζοντας την θέση των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο. Ένα ιστορική σημασία βήμα προς τα εμπρό όσον αφορά το Κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια για την Σερβία δεν αναγνωρίζεται η ίδια η ανεξαρτησία στο Πέδιο, αλλά αναγνωρίζεται η πραγματικότητα επιτόπου στο Πέδιο και η πραγματικότητα για την, ε, τις ανάγκες που έχουν οι Σέρβοι στο Πέδιο λαμβάνονται έτσι υπόψη. Με αυτή τη συμφωνία συμφωνήθηκε ότι η κοινότητα των ε, δήμων των ε, Σέρβων στην ε, περιοχή Κωσυφοπεδίου Μετόχια θα διέπεται από την αρχή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων όσον αφορά τα δικαιώματα, την χάρτα δικαιωμάτων αυτών των κοινοτήτων σε σχέση με την σερβική μειονότητα τα θεσμικά όργανα στο Κωσυφοπαίδιο και την Μετόχεια θα εποπτεύονται από την Πρίστινα, αλλά με σαφή δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα αυτονομίας αυτής της σερβικής κοινότητας και όσον αφορά την δράση της και όσον αφορά και την χρηματοδότηση των δικαιωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει μια ξεχωριστή δημιουργία μιας ξεχωριστής δημοκρατίας των Σέρβων, διότι αυτό δεν είναι ο στόχος. Νομίζω όμως ότι αυτή η συμφωνία είναι μια, ένα νέο βήμα σε μια νέα σχέση μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας για τη διασφάλιση της, ε, ενός πλαισίου ασφάλειας υπέρ όλων των κοινοτήτων και θα αποτελεί την βάση για μια πολύ ε, επιταχυμένη νέα οικονομική ανάπτυξη. Το αναγκαίο επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός ημερομηνία για την έναρξη διαπραγματεύσεων και η προϋπόθεση είναι η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας με την Πρίστινα. Πρόθεσή μας είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία συμφωνήσαμε με την ε, Πρίστινα του Κωσυφοπεδίου και δεν υπάρχει κανένα δίλημα σχετικά με αυτά. Η Σερβία υλοποίησε το σχέδιο, ενέκρινε το σχέδιο ε, δράσης ε, για αυτή τη συμφωνία και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της η σερβική κυβέρνηση για να υλοποιηθεί πλήρως αυτή η συμφωνία και να έρθουν τα προσκόμματα και τα εμπόδια, τα τελευταία εμπόδια τα οποία υπάρχουν ώστε να ληφθεί απόφαση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για ημερομηνία έναξης διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στι μεταρρυθμίσεις που έχουν ε, προχωρήσει στην Σερβία. Εμπλεκόμεθα ως κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού κλάδου. Ε, και όσον αφορά το, ε, τη δικαστική εξουσία έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για τη λειτουργία της Δικαστικής Ακαδημίας και το πρόγραμμα δράσης ε, για τα επόμενα πέντε έτη. Ο κύριος στόχος είναι να εγκριθεί ένα διαφανές δικαστικό σύστημα το οποίο θα προάγει το κράτος δικαίου και την, τα θέματα δικαιοσύνης η καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να αξιολογηθεί ως μια πολύ θετική δράση. Αναγνωρίστηκε αυτό στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντάχθηκε σε σχέση με τη Σερβία. Η έγκριση μιας νέας στρατηγικής και μιας νέας ε, δράσης κατά της διαφθοράς ε, πρόκειται να εγκριθούν και η μηδενική ανοχή μας έναντι της διαφθοράς ε, και η επιβολή κράτους δικαίου είναι στόχοι μας. Επίσης η επόπτευση των μηχανισμών σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ αυτών και μεταξύ της, ε, των αστυνομικών αρχών και των διοκτικών αρχών θα ήθελα να τονίσω πέρα από το γεγονός ότι κατά τα τέλη του 2012 τροποποιήσαμε το νομοθετικό μας πλαίσιο και κάποιες διατάξεις νομοθετικές. Για εφέτος το 2013 θα έχουμε πιο εξειδικευμένες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ε, του ποινικού κώδικα που θα δημιουργήσουν την ε, ραχοκοκαλιά για τη δράση μας κατά της διαφθοράς. Ευρίσκεται καθοδόν η στρατηγική για την μη διακριτική μεταχείριση και έχουμε υπόψη την προαγωγή και υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγική μας ε, θα ε, βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά τις ε, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα βελτιώσει την θέση τους. Μέτρα και διαβήματα έχουν αναλυθεί για την ενίσχυση των ετούντων άσυλο και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τα τέλη του 2012 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των ετούντων άσυλο και το παράδειγμα της Γερμανίας δείχνει ότι μειώθηκαν σημαντικά οι αριθμοί ετούντων άσυλο που προέρχονται από την Σερβία ή πέρασαν από τη Σερβία στην ε, Γερμανία και ζήτησαν άσυλο. Ανταποκρινόμαστε στις προδιαγραφές και απαιτήσει. Είναι αναγκαίο όμως ε, να καταργηθεί το καθεστώς ε, θεωρήσεων διαβατηρίων που έχει αρνητικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα μειονοτικά δικαιώματα, η κυβέρνησή μας ενεργά δραστηριοποιείται για να εγκριθεί και να υλοποιηθεί μια νέα στρατηγική προσέγγιση. Θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους ευάλωτους, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ευάλωτες μειονοτικές ομάδες ε, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αρνητική διακριτική μεταχείριση. Θα υπάρξουν κύρια άξονες για τη δράση μας ε, όσον αφορά τους άξονες αυτούς, ε, λαμβάνοντας ολοκληρωμένα μέτρα για την βελτίωση της κοινωνικής θέσης αυτών των ομάδων και της κατάργησης της αρνητικής μεταχείρισης. Όσον αφορά τις μειονότητες, πρόοδος σημειώθηκε κατά την τελευταία περίοδο, ιδιαίτερα με μια πιο τακτική βάση με το Συμβούλιο των Εθνικών Μειονοτήτων. Άρθηκαν εμπόδια όσον αφορά την χρηματοδότηση μειονοτήτων και πρωτοβουλίε αναλύθηκαν ώστε να επαναδραστηριοποιηθούν οι, ε, οι δυνατότητε των ε, μειονοτήτων αυτών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα πιο σημαντικά θέματα που είναι ε, η οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα που απορρέουν από την οικονομική κρίση στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσμια κλίμακα. Τα προβλήματα αυτά είχαν σημαντικότατες επιπτώσεις ε, στη Σερβία και η αύξηση της ανεργίας που έχει ξεπεράσει τα 25% είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο μισθών και αμοιβών. Ε, η ε, μείωση του βιωτικού, η υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών μας είναι ανησυχητικό επίπεδο. Παρότι υπάρχουν και ενθαρρυντικά στοιχεία ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες η Σερβία που μπορεί να δώσουν θετικές προοπτικές. Ιδιαίτερα η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις στη Σερβία δείχνοντας ότι θα υπάρχουν πλεονεκτήματα για τέτοιες ε, ε, επενδύσεις μια και θα υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα υπέρ αυτών. Το σύστημα φορολόγησης ε, και η μικρότερη φορολόγηση και το σύστημα προτιμήσεων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις, συνεργασία επιπλέον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με το, την κοινοβουλευτική συνέλευση της Δημοκρατίας τη Σερβία, μέσω ενός κοινοβουλευτικού διαλόγου η αντιπροσωπεία της Σερβικής Βουλής σε σχέση με τις την αντιπροσωπεία για τις νοτιοανατολικοευρωπαϊκές χώρες και το ε, ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικά φόρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε ότι με την επόμενη σύνοδο κορυφής θα αναβαθμιστούν οι σχέσεις ε, αυτών των θεσμικών οργάνων και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν επαφές που θα καλλιεργηθούν με τους ομολόγους και εταίρους μας. Η υποστήριξή σας για την προοπτική ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σημασία. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό όπω και η οικονομική ανάπτυξη τη Σερβία για την περιοχή τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτό είναι η πολιτική διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω πρωθυπουργό ε, αυτή τη χώρα, ε, μια χώρα ε, που έχει εμπορικέ σχέσει με τις ευρωπαϊκές χώρες σε επίπεδο των δύο τρίτων των ε, συναλλαγών μας. Θέλω να απευθύνω έκκληση να δοθεί συνέχεια στην προοπτική διεύρυνση. Δεν πρέπει να επιβραδυνθεί μετά την πρόσβαση της ε, ε, Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτό τα οποία, τα οποία αντιμετωπίζει η Σερβία και η πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις πιο επιτυχείς ευρωπαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα. Σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών αναβαθμίστηκαν και βελτιώθηκαν και βρίσκονται όλα αυτά στον πυρήνα της ύπαρξης και δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της, του μεγαλύτερου πολιτικού εγχειρήματος υπέρ της, ειρήνευσης, της ειρήνης στην Ευρώπη η Σερβία δεν ζητεί να υπάρξουν, να ξεχωριστοί κανόνες και ρυθμίσεις για αυτήν, αλλά αυτά τα οποία είναι γνωστά και αναγνωρισμένα ως τα κριτήρια για ένταξη άλλων κρατών μελών πρέπει να εφαρμόζονται και για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας διασφαλίζω ότι από πλευρά της η Σερβία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ανταποκριθεί. Η πορεία για την ένταξη της Σερβίας έχει κέρια σημασία για την ολοκλήρωση της ευρύτερης περιοχής και την ε, ευρωπαϊκή της προοπτική. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες που κατέβαλε η προσπάθεια με τέτοιο τρόπο ώστε η Σερβία και η συνολική ευρύτερη περιφέρεια να προσεγγίσει περισσότερο πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθεί η ευρωπαϊκή προοπτική και κάποτε να γίνουμε δεκτοί ως πλήρη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κατακλείδη πολύ για την υποστήριξη που προέρχεται από μεγάλο αριθμό ευρωβουλευτών και σας ευχαριστούμε και για την υποστήριξη να γίνει το Βελιγράδι το 2020 πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι για μας αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων Επίσης, λόγω του ότι υπάρχει εδώ το συγκεκριμένο στοιχείο των διαφορετικών πολιτικών επιρροών ε, της μεγάλης πολιτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς της Σερβίας ιστορικά που ήταν μια χώρα που επί πάρα πολλά χρόνια βρισκόταν στο μετέχμιο μεταξύ του ρήγματο που χώριζε την Δύση από την Ανατολή. Μια χώρα στην οποία γεννήθηκαν πολλοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες, μεταξύ άλλων και ο μεγάλος Κωνσταντίνος που κάπου 17 αιώνες πριν ενέκρινε το διάταγμα των Μεδιολάνων με το οποίο νομιμοποιήθηκε, νομοθετήθηκε η χριστιανική θρησκεία στην Ευρώπη και έγινε επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είμαι στη διάθεσή σας όπως ανέφερα, στον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Εξωτερικών για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις θα είχατε και να ακούσω όλες σας τις προτάσεις. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι έχασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Σερβία μέχρι σήμερα. Το ΑΕΠ της Σερβίας είναι 65% εκείνου που ήταν το 1989 έχει μειωθεί σημαντικά. Η Σερβία δεν μπορεί να κάνει μικρά βήματα προς τα εμπρός. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι άλματα, αυθεντικά άλματα για να σημειωθεί πρόοδος. Ακριβώς επειδή το έθνος μας, οι πολίτες μας ε, βιώνουν τα πάνδυνα σήμερα και αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Πρέπει όλα αυτά μέσα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία η πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι το πιο δύσκολο πάντα. Εμείς πιστεύουμε ότι ήδη κάναμε αυτό το πρώτο πιο δύσκολο βήμα και επιτρέψτε μου να σας διασφαλίσω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη, ιδιαίτερη υπευθυνότητα θα δράσουμε στο, στα όσα έχουν συμφωνηθεί με την Πρίστινα στο Κωσυφοπέδιο και για τις εσωτερικές μας μεταρρυθμίσεις στη Σερβία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό καλωσόριμα στον κύριο Τάτιτσε, τον Πρωθυπουργό. Χαιρόμαστε που ήρθατε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Γνωρίζω λιγάκι τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή και γνωρίζω πολύ καλά ότι με τις αλλαγές που εισαγάγατε, με αυτές τις αλλαγές επιδείξατε μεγάλο προσωπικό και πολιτικό θάρρος. Τα αποτελέσματα που έχει να επιδείξει η νέα κυβέρνηση της Σερβίας είναι ενθαρρυντικά. Θυμάμαι παλαιότερα το πρόγραμμα με βάση το οποίο σχηματίστηκε ο συνασπισμός ανέφερε με απόλυτη σαφήνεια ότι επιθυμείτε να ακολουθήσετε τον ευρωπαϊκό δρόμο. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μέχρι τώρα τηρείτε αυτά τα οποία έχετε πει και έχετε και στοιχεία να τεκμηριώσετε αυτή σας την άποψη. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή έχετε προχωρήσει τόσο πολύ σε αυτό το δρόμο, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε. Ξέρω πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος αυτός. Νομίζω όμως ότι ε, έχετε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη όλων μας. Επίσης ε, θέλω ε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη των μελών ε, της αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη για το γεγονός ότι όταν επισκεφτήκαμε το Βελιγράδι ήσασταν στη διάθεσή μας όχι για πέντε λεπτά αλλά για δύο ώρες και μάλιστα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ώρες. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι με τις συζητήσεις που είχαμε και προσβλέπουμε να ξανασυναντηθούμε είτε εδώ είτε στη Σερβία. Η ιστορική αλλαγή της ε, Σερβίας και η στροφή της ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και είναι ένα Ηράκλειο καθήκον. Αλλά αποδείξατε ότι είσαστε αποφασισμένος να προχωρήσετε και ακολουθείτε με συνέπεια αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν ε, μπορείτε να έχετε την εμπιστοσύνη όλων μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν απόλυτα κατανοητές και επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση για να μπορέσετε κι εσείς ε, να εκφράσετε τις απόψεις σας για ένα θέμα που κατά την άποψή μου ε, λανθασμένα προκαλεί ανησυχίες στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τις σχέσεις Σερβίας και Ρωσίας. Ορισμένοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι στην ε, πολιτική σας ε, εντοπίζει κανείς ένα έντονο φιλορωσικό στοιχείο. Και πολλοί ε, το επικρίνουν αυτό. Το να έχει κανείς καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αυτό δεν είναι κακό, όλοι το επιθυμούν. Και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι. Όμως στη δική σας την περίπτωση υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες επ' αυτού. Υπάρχουν ε, ιστορικοί δεσμοί Σερβίας και Ρωσίας και καλών σχέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μας εξηγήσετε λιγάκι την στάση σας και τις απόψεις σας και αυτό για να μην υπάρχει τροφή για περιττές εικασίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, συνάδελφοι, έχω ένα μακρύ κατάλογο ε, θα έχουν όλοι από δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριος Κατσίν. Θα ήθελα να πω το εξής. Σας ε, καλωσορίζουμε καταρχήν εδώ. Η επίσκεψή σας ε, δείχνει ότι επιθυμείτε να συνεχίσετε το δρόμο της ευρωπαϊκής ένταξης. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τις ε, προσπάθειες ε, της κυβέρνησής σας έτσι ώστε να αποκτήσετε ημερομηνία έναρξης ε, διαπραγματεύσεων. Η επίσκεψή σας εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ενθαρρυντική για όλους μας. Πρέπει να εξηγήσετε στους συναντέλφους γιατί αξίζει στη Σερβία να πάρει την ημερομηνία. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι με την επίσκεψή σας εδώ μπορείτε να διευκολύνετε το καθήκον μας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι ο ρόλος της ε, Σερβίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να το μιμηθούν χώρες όπως η Μακεδονία, η Βοσνία Ερσεγοβίνη, δείξατε πώς ε, η Σερβία, πώς ε, μια χώρα μπορεί να ακολουθήσει μια ρεαλιστική πολιτική. Πώς αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειές σας πρέπει να επενεθούν και πρέπει να μελετήσει κανείς την Ευρώπη αλλά και αλλού τις ε, σχέσεις με τον κύριο Ντάτσι όπου υπάρχουν εκρεμείς διαφωνίες. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά την εφαρμογή, τι ακριβώς προτίθεστε να θέσετε σε εφαρμογή στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Το θέμα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία, ε, Ιούνιος. Τι έχετε συμφωνήσει από αυτού. Και τέλος, στα μέσα ενημέρωση της Σερβίας αναφέρεται σήμερα ότι πρόκειται να υπάρξει ανασχηματισμός της κυβέρνησής σας. Για ποιον ακριβώς λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ ε, όσον αφορά αυτό το ιστορικό βήμα που κάνατε να υπογράψετε την ιστορική συμφωνία με το Κοσμοπέδιο γιατί με αυτόν τον τρόπο επουλώνονται οι πληγές και αποκαθίστανται οι αδικίες. Είναι πολύ σημαντικό να καταδικάζει κανείς τη βία και τη μυσαλλοδοξία και ε, παλαιότερες προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο πρέπει πράγματι να προχωρά κανείς. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα με την ευκαιρία που ήρθατε εδώ να σας ε, κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζω και θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι στα μέσα ενημέρωσης, ε, στις ε, μετακομμουνιστικές χώρες ε, μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία της Ιουγκοσλαβίας, της πάλε ποτέ Ιουγκοσλαβίας. Θα πρέπει να ε, προσφέρονται τα αρχεία αυτά στις ε, ανεξάρτητες δημοκρατίες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο στη Σερβία και αλλού, λόγω του ότι υπήρχε αυτό το σύστημα των πρακτόρων ε, στο οποίο είχαν ε, ενταχθεί διπλωμάτες, ε, κληρικοί. Περίπου η ίδια κατάσταση είναι και στη και μου τη χώρα, τη Βουλγαρία. Εσείς, τι πιστεύετε από αυτού. Τάσεστε υπέρ του να ανοίξουν τα αρχεία ή όχι. Η εμπειρία δείχνει ότι οι νεόκοπες δημοκρατίες που ακολούθησαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και έδειξαν αυτή την τόλμη, αυτό το θάρρος να ανοίξουν τα αρχεία τους, τα πήγανε πολύ καλύτερα από τις άλλες ε, που τα κράτησαν απόρριτα. Και εύχομαι πραγματικά καλή τύχη στη Σερβία, στον δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Μπορείτε να βασιστείτε στη δική μας την υποστήριξη. Ευχαριστούμε τώρα ο κύριος Βάλτσακ, πρόεδρος της Ομάδα Εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Πρωθυπουργέ. Πρώτα απ' όλα να σα συγχαρώ για την τόλμη σα. Διότι ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να ασχολείται κανεί με θέματα τόσο ακαθόδη και ευαίσθητα από ιστορική πολιτιστική και πολιτική άποψη. όπως ε, το κοσφοπέδιο και, και τα μετόχια. Σας ε, συγχαίρω λοιπόν για τις προσπάθειές σας και την υλοποίηση όλων των συμφωνημένων. Εμείς ως ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εκτιμούμε και τις προσπάθειές σας για μεταρρυθμίσεις. Αναφέρατε όσα γίνονται για τις εθνοτικές μειονότητες και το κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Και ακριβώς θα πρέπει να ανταμυφθείτε για αυτές τις προσπάθειες. Τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της, οι κυβερνήσει των κρατών μελών να παραμείνουν πιστοί στι υποσχέσει του. Και στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα τη Σερβία. Αυτή είναι η δική μα επίσημη θέση. Αναφέρατε το έτος 2020, πόσο σημαντικό θα είναι για το Βελιγράδι. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή την ημερομηνία να την έχουμε λίγο πολύ στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν συζητούμε περί διεύρυνσης και όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Όχι μόνο για το Βελιγράδι, για ολόκληρη τη Σερβία. Η Σερβία είναι μια ζωτική σημασία χώρα, ένα στρατηγικό παράγοντα για όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Και θέλω με αυτό να έρθω και στην ερώτησή μου. Μιλήσατε για την οικονομία. Ξέρουμε πόσο δυσχερεί είναι οι συνθήκε αυτή τη στιγμή. Έχετε 20% ανεργία και ακόμα μεγαλύτερα για τους νέους ποσοστά. Ε, χρειάζονται λοιπόν στρατηγικά προγράμματα για τις υποδομές. Και εδώ έχω στο μυαλό μου το εξής. Αυτοκινητόδρομους και τρένα ταχείας κυκλοφορίας. Διασύνδεση του Βελιγραδίου λοιπόν με τις κοντινές πρωτεύουσες Βουδαπέστη, Βουκουρέστη, Σόφια. Αυτό δεν θα μπορούσε ως ε, εγχείρημα να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστούμε κυρία Μπέντνερ. Ευχαριστώ θερμά. Θερμά καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ πράγματι για αυτά τα οποία εσείς με μεγάλο θάρρος και μεγάλα, ε, μεγάλο όραμα, μακροπρόθεσμο όραμα υλοποιήσατε. Δηλαδή μακροπρόθεσμα να μπορέσετε να οδηγήσετε την πορεία της Σερβίας ε, είναι κάτι το οποίο καλοχαιρετίζουμε και σας συγχαίρουμε για αυτή την πρωτοβουλία σας και κυρίως και περαιτέρω ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η πορεία σας προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου δύο σύντομε ερωτήσεις και ένα σχόλιο. Μία ερώτηση, τι σκέπτεστε να πράξετε ώστε οι Σέρβοι στο βόρειο Κωσυφοπέδιο να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Δηλαδή να προσελκύσετε τους Σέρβους αυτούς να δείξουν κατανόηση σε αυτά τα οποία σχεδιάζεται. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Πολλά μπορούν να υλοποιηθούν αν οι άνθρωποι επιτόπου όμως δεν συμμετάσχουν δυσχεραίνονται τα πράγματα. Γι' αυτό ανεξάρτητα από τα βήματα υλοποίησης Ποια είναι η δική σας, ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός και τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να ε, προσελκύσετε τους Σέρβους να συμμετάσχουν. Και μετά σε σχέση με την ε, ολοκλήρωση, σε σχέση με τις ε, αρχές, τι θα γίνει ώστε και σε σχέση με τα επιμέρουσα άτομα να μπορέσετε να προχωρήσετε στην δημιουργία των αστυνομικών αυτών δυνάμεων σε σχέση με την αφήνιση των ρόλων, τι θα μπορούσατε να πείτε ότι μπορεί να προχωρήσει. Και ένα τελευταίο σημείο. Προηγούμενα αναφερθήκατε στην οικονομική κατάσταση της Σερβίας και στο ότι βλέπετε το φως στο τέλος της σύραγγας, στην άκρη της σύραγγας βρίσκεστε ακόμα σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση και τα πρόσφατα στοιχεία όσον αφορά το ε, Χρηματοδοτικό Συμβούλιο είναι ανησυχητικά και γίνεται έκκληση και ζητείτε να αναλυθεί μεγαλύτερη δράση και μέσα σε αυτή την συγκυρία πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ελαφρά την καρδία να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα στοιχεία. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι στην ε, Γερμανία θα δώσουμε μάχη για την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευρά ε, τη ε, Γερμανία είμαστε υπέρ μια ε, μεγαλύτερη ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να υπαρκεστούμε με την ένταξη τη Κροατία. Πρέπει να ακολουθήσει η Σερβία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάνοκ, παρακαλώ. E Καλώ ήρθατε κύριε Ντάτσιτ από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Είμαι φίλο τη Σερβία και καλωσορίζω την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Οι προτάσεις μου και οι προβλέψεις για μια σωστή ε, διέρεση ίσως να είναι πλέον περίτη ε, και να βρεθεί μια καλύτερη λύση. Όμως, ξέρουμε ότι μέλη της κυβέρνησής σας έχουν ευχαριστεί από τα πλήθη γιατί κάποια από τα εθνικιστικότερα στελέχη έχουν ε, δεχτεί φοβερά επικριτικά σχόλια. Αυτό πώς αντιμετωπίσετε. Χθε ήταν παρόν και ο κύριος Κούκαν και μας είπε ένας εκπρόσωπος από τη Βοσνία και Ζεγοβίνη, ότι δεν μπορούμε τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να τους αφήσουμε τελείως στην τύχη τους. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι και οι δικές, τα δικά του συμφέροντα μπορούν να καλυφθούν μακροπρόθεσμα με έναν τρόπο διορατικό. Δηλαδή το τι θα γίνει και με τη Μητρόβιτσα και τις κοινότητες Σέρβων ε, εκεί. Ο κύριος Κούκαν ρώτησε για τις σχέσεις σας με τη Ρωσία. Μπορώ να σας ρωτήσω τι γίνεται και με τους ε, γείτονες, όπως με το Μαυροβούνιο. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων ε, για το Μαυροβούνιο και την προσχώρησή του στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μπορείτε να προλάβετε τι εξελίξει στο Μαυροβούνιο και να προσχωρήσετε ταυτόχρονα. Και τι βλέπετε να γίνεται με τη Μακεδονία που τα πράγματα έχουν καθυστερήσει και δεν υπάρχουν πλέον συνομιλίε και διαπραγματεύσει. Τι θα γίνει με το θέμα τη ονομασία. Και ένα τελευταίο ευαίσθητο θέμα. Ε, η Κροατία πρόκειται να προσχωρήσει και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Όμω πιστεύετε ότι κινδυνεύει να δυσκολεύσει τη σα διαδικασία προσχώρηση η λόγω τη προδεκαετία σύγκρουση που υπήρξε μεταξύ σα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τζαβέλα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώ ήρθατε. Είναι τιμή μα και προνόμιο να σα έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Σα ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και για τη Σερβία και για την ευρύτερη περιοχή η έναρξη διαπραγματεύσεων με επίσημη ημερομηνία για τη Σερβία θα σημαίνει το τέλο μια μακρά περίοδου αστάθεια για την περιοχή. Η δική μου ερώτηση είναι η εξή. Τι άμεση περιφερειακή συνεργασία και σχετικέ πρωτοβουλίε αναμένεται να ε, αναλυθούν. Πώ θα θέλατε οι γειτονικέ σα χώρε να αξιοποιήσουν αυτή την ιστορική ευκαιρία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, με μεγάλη χαρά σας ε, βλέπουμε σήμερα εδώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να διοργανώνουμε διασκέψεις για τους φίλους της Σερβίας ε, με τους διάφορους εκπροσώπους. Θα πέρασω στα ρουμανικά. Άστο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας πω το εξή ε, και να το πω και προς τους συναδέλφους. Μόνο εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν την τεράστια περιπλοκότητα αυτής της κατάστασης γνωρίζουν και τις τεράστιες ευθύνες που επομίζεστε και μέσα σε αυτό αυτή την προοπτική, το τεράστιο θάρρος το οποίο εσείς ε, απαιτείτε να δείξετε και καταδείξατε στην ε, Πρίστινα και στο Βελιγράδι και κάνατε αυτό το ιστορική σημασία βήμα. Σας παρακαλώ λοιπόν τα πολιτικά κόμματα να γνωστοποιήσετε σε αυτά στο Βελιγράδι ότι γνωρίζουμε να αξιολογήσουμε σωστά πώς ε, αυτά πρέπει να αξιολογηθούν αυτά τα βήματα τι κάνατε δηλαδή ώστε η μειονότητα η σερβική να αποκτήσει αυτή την προοπτική. Είναι ένα ιστορικό βήμα. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι μπορούν τα πράγματα να εξεταστούν και υπό διαφορετική προοπτική. Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξουν για τη Σερβία νέοι όροι και προϋποθέσεις που θα προσθεθούν στην ε, αξιολόγησή της. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο θα καθορίσει μια ημερομηνία για την έναξη των ε, διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων για την ε, προσχώρηση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό επειδή ο ρόλος της Σερβίας για την περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ουσιώδης, είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο ρόλος της Σερβίας Γνωρίζουμε να αξιολογήσουμε αυτά τα πράγματα και τα τεκτενόμενα από πλευρά της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, θα μου επιτρέψετε βεβαίως ε, να μιλήσω σλοβενικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεταρρύθμιση της πολιτικής σας και για την πολιτική επί της οποίας συμφωνήσατε με τον εταίρο σας στην κυβέρνηση συνασπισμού. Πρόκειται για μια σύγχρονη πολιτική, μια πολιτική που ε, αντικατοπτρίζει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δρόμο. Παλαιότερα εμείς προετοιμάζαμε ένα ε, χρονοδιάγραμμα και ένα χάρτη πορείας για το κοσφοπέδιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χάρτη πορείας ε, ε, πλέον συμπεριλαμβάνεται στις σχέσεις από τις οποίες έχετε συμφωνήσει. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Η Σερβία και δικαίως έχει καταλήξει μια νέα πολιτική γραμμή και ελπίζω ότι θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χαιρόμουν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και έχω να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά στις πολιτικές δραστηριότητες, σχετικά με την αυτονομία της Βοηβοντίνα, εντάσσονται αυτές στη δική σας την πολιτική ή θα αφήσετε τη Βοηβοντίνα να είναι απλά ένα στοιχείο πρωτοπόρου πολιτικής. Ε, όσον αφορά τις, ε, τους πρώην δήμους ε, στα βόρεια του Κοσμοπεδίου, δεν πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει το σύστημα και τη σχέση με την οποία έχετε, για την οποία έχετε συμφωνήσει με την Πρίστινα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και ελπίζω να μπορέσετε να πείσετε την κοινή γνώμη ότι η πολιτική σας ε, θα στεφτεί από επιτυχία και ότι θα τολμήσετε να κάνετε τα βήματα που χρειάζονται. Κυρία Κοπά, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας έχουμε εδώ ενώπιον μας. Ως χιώτης εισηγήτρια για τη Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα για τη Σερβία, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την θετική σας θέση και στάση όσον αφορά την αντιμετώπιση του κοσυφοπεδίου και όπως πολλοί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους ανέφεραν, αυτό είναι ένα υπόδειγμα και θα έπρεπε να είναι ένα παράδειγμα και για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν περιφερειακές τέτοιες αντιπαραθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα λοιπόν άλλο πλέον προς σχηματικά και πρέπει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει ε, για την ένταξη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική μα ομάδα θα σα υποστηρίξει σε όλε σα τι προσπάθειες ε, που αφορούν τι μεταρρυθμίσει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την ε, σερβική κυβέρνηση σε πολλού τομείς. Αλλά όσον αφορά την, το Ευρωκοινοβούλιο θα μας βρείτε στο πλευρό σας σε αυτή την προσπάθεια. Όπως πολλοί από τους συναδέλφους έθεσαν ερωτήματα για τις σχέσεις σας με διάφορες χώρες εγώ θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τις σχέσεις μεταξύ της Σερβίας και την Τουρκία που είναι σημαντικός περιφερειακός ε, εμπλεκόμενος ε, ως δύναμη. Γνωρίζουμε ότι σε σχέση με τις στενότερες αυτές σχέσεις με την Τουρκία θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη ποια είναι. Ευχαριστώ. Κυρία Λούνατσεκ παρακαλώ. Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και εκ μέρου των Πρασίνων να σα καλωσορίσω και εγώ εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επειδή και εγώ είμαι συγκήτρια για το κοσμοπέδιο, ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για όσα εσεί, και η κυβέρνησή σα έχετε κάνει από τότε που αναλάβετε την εξουσία πέρσι. Όταν συναντήκαμε πέρσι, πριν ακόμη αναλάβετε τα ενία, η δέσμευσή σα τότε, οι υποσχέσει σα μα είχαν εντυπωσιάσει. Όπω είπε ο συνάδελφο Κούκαν, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσωπική σας δέσμευση, για την πολιτική σας τόλμη και πυγμή να αναλάβετε αυτό τον μαραθώνιο, αυτό τον άθλο που ξεκινήσατε από πέρσι. Έχετε φτάσει κοντά στο τέρμα των 40 χιλιόμετρων και μένουν περίπου 2-3 ε, για να ολοκληρωθεί ο δρόμος, ε, να κλείσει η κούρσα. Ε, Ξεκίνησατε πέρσι και ελπίζω πραγματικά ότι θα πετύχετε και ότι θα τελειώσει η διαδρομή. Ε, ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία Σερβία-Κωσυφοπεδίου και ότι επιτέλου θα έχετε μια ημερομηνία, επίσημη ημερομηνία για την άνοιξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρησή σα. Ελπίζουμε ότι και το ε, θα υπάρξει και μια συμφωνία σύνδεση και συνεργασία και με το κοσμοπεδίο. Ε, Όπω σε κάθε μαραθώνιο βεβαίω υπάρχουν ε, ακόμη κάποια μικρά εμπόδια. Θα ήθελα λοιπόν ένα-δυο στοιχεία τα οποία πρόσφατα αντιλήφθηκα να σα σχολιάσω. Το Σαββατοκυριακό θα υπάρξει μια σύνοδο τη διαδικασία συνεργασία με την Ανατολική Ευρώπη και με ε, εκπροσώπου υψηλού επίπεδου καθώ και με τη συμμετοχή υπουργών και πρωθυπουργών. Ε, άκουσα ότι δυστυχώ Ακόμη και εφόσον απεστάλλει πρόσκληση στο, από το ΕΣΥ στον πρόεδρο του Κοσμοπεδίου, ότι η συμμετοχή αυτή δεν θα γίνει, δεν θα υπάρξει από τον πρόεδρο Νίκολίτ. Και μάλιστα άκουσα ότι κάποιες από τις πρεσβείες σας δεν ευθυγραμμίζονται ακόμη με την συμφωνία που έχετε εκφράσει. Ότι κάποιοι συμμετέχουν σε συναντήσεις, σε διασκέψεις ενεργά στη χώρα σας, τι θα κάνετε λοιπόν ώστε όλοι, με συγχωρείτε, όλες οι σερβικές αρχές, όλοι οι επίσημοι φορείς και εκπρόσωποι της Σερβίας να ευθυγραμμιστούν μας αποφασίσετε σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τη χώρα σας αν θέλετε να προχωρήσουμε ε, και να έχετε την πλήρη στήριξή μας. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα ο κύριος Μιρέλα από την Γενική Διεύθυνση Διεύθυνσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου τιμή να μπορώ να εκφράσω και εγώ την δική μας εκτίμηση για τις ε, ιστορικές προσπάθειες της Σερβίας, για να το πω έτσι. Και εσάς προσωπικός Πρωθυπουργέ, για το όραμα που βλέπουμε ότι επιδιώκεται να υλοποιήσετε όλους τους περασμένους μήνες τον διάλογο ψηλού επίπεδου με το Κοσμοπέδιο, όπω διευκολύνθηκε από την είπατε εκπρόσωπο τη Λέδη Άστον. Μια θεώρηση που με τα δικά σας λόγια ε, ήταν ε, κάτι που εμπνευστήκατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Αυτό το είπατε και εσείς στις εναρκτήριες παρατηρήσεις σας. Ε, η ενεργό σας συμμετοχή στο διάλογο και οι τολμηρές κινήσεις που κάνατε. Κάτι που και στη χώρα σας προβλήθηκε σωστά είναι κάτι που είναι αξιοέπαινο. Πραγματικά Έχουμε ήδη αποσπάσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, για το μέλλον της πορείας του κοσφοπεδίου Θέλουμε μια σταθερή υλοποίηση του προγράμματος δράσης καθώς και των υπολείπων στοιχεία, στοιχείων που έχουν ε, ήδη συμφωνηθεί και ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα για τα ενεργειακά και τις τηλεπικοινωνίες η κίνησή σας προς το κοσυφοπαίδιο είναι σημαντικότατη και για τους πολίτες και στις δύο πλευρές αλλά και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ως ε, θετικό παράδειγμα να αναφέρω μάλλον ότι ο αριθμός ε, των διμερών θεμάτων, των θεμάτων που διμερώς πρέπει να συζητηθούν στην περιοχή και κρεμούν, είναι ακόμα σημαντικός, αλλά ο Επίτροπος Φίλε πρόσφατα επισκέφθηκε την ε, χώρα και είπε ότι η κυβέρνησή σας έχει αναλάβει δράση και αναμένεται οι στρατηγικές στους τομείς ε, των δικαστικών, την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, την μη διακριτική μεταχείριση. Όλα αυτά τείνουν να ευθυγραμμιστούν με τις δικές μας συστάσεις. Και αυτά σήμερα είναι σημαντικότατα στοιχεία όπως ε, υπενθύμησε ο πρόεδρος μας, ο, κύριος, ο πρόεδρος ο κύριος Μπρόκ μάλλον. Εδώ συμμεριζόμαστε τις ε, υψηλές φιλοδοξίες που εξέφρασαν πολλοί από τους βουλευτές σήμερα το πρωί, ότι η Σερβία θα προσκληθεί επιτέλους στα τέλη Ιουνίου να περάσει στην επόμενη φάση να ξεκινήσει την επίσημη πορεία της προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πολλές, πολλαπλές ερωτήσεις. Μπορείτε τώρα να απαντήσετε. Ευχαριστώ θερμά κυρίες και κύριοι αγαπητοί ευρωβουλευτές. Οι ερωτήσεις αυτές ε, είναι πολύ πιο εύκολο να απαντηθούν από εκείνες τις οποίες θα πρέπει να απαντήσω στο Σερβικό Κοινοβούλιο υστερότερα, διότι θα έχουμε και οικονομικά θέματα ε, που εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που παρενέβησαν και για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνεται όσον αφορά την κατάσταση στη Σερβία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα ενθαρρυντικά λόγια και λόγια υποστήριξης που εκφράσατε για τα όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε και τις προσπάθειές μας. Οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν αφορούν κάποια θέματα στα οποία τοποθετήθηκα ή απάντησα ήδη, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Υλοποίηση, εφαρμογή. Συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα υλοποίηση για την εφαρμογή του. Καθορίζει ημερομηνίε, διορίες, ε, πράγματα, κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό το σχέδιο αποτελείται από διάφορα τμήματα. Πρώτον, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου θεμελιώδους σημασίας για την εφαρμογή της συμφωνίας που πρέπει να γίνουν όλα αυτά από τις δύο πλευρές αμφωτέρωθεν. Έχουμε και το θέμα του δικαστικού, της δικαστικής εξουσίας και τις τοπικές εκλογές το φθινόπωρο, δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν, την λειτουργία της κοινότητας των Σέρβων, των κοινοτήτων των Σέρβων μέχρι ότου γίνουν αυτές οι εκλογές θα πρέπει να συνέλθουν οι ομάδες εργασίας στο εγγύς μέλλον και αναμένουμε ότι με τη, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ή οι παρόλες τις ευρύτερες πιέσεις ε, το σχέδιο αυτό θα μπορέσει να υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Τώρα, σε σχέση και παράλληλα με το σχέδιο αυτό για την ε, εφαρμογή του συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις για τα ενεργειακά θέματα και τις τηλεπικοινωνίες. Και εδώ επίσης υπάρχουν διορίες ε, που πρέπει να επιτευχθούν. Και αυτά τα θέματα είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Και θα πρέπει επίσης να επενδύσουμε και πολλά να πράξουμε, πολλές προσπάθειες να καταβάλουμε για να επιτευχθεί ένα συμβιβασμός είχαμε μια πολύ σαφή συγκεκριμένη προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Δεν συζητήσαμε θέματα καθεστώτος. Ε, ο διάλογος αφορούσε συνολικά ευρύτερα θέματα και σε σχέση και με την αναγνώριση του ζητήματος αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου από τη Σερβία ως ζήτημα δεχτήκαμε να συζητήσουμε το θέμα του κοσυφοπεδίου με βάση το ψήφισμα 12-11 των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμετοχή των Σέρβων στην πολιτική ζωή, στο πολιτικό γίγνεσθε του κοσυφοπεδίου και αυτό συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών και τροποποιήσεων σε σχέση με τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα, την δημιουργία και νέων θεσμικών οργάνων επιπλέον όσον αφορά και την υλοποίηση στη συνέχεια της ε, συμφωνίας αυτής. Είναι προς το συμφέρον μας οι Σέρβοι στο, βόρειο του, στο βορρά του Κωσυφοπεδίου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση, την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως η συμφωνία αυτή αν εφαρμοστεί μόνο από το Βελιγράδι χωρίς αυτούς. Και γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί ένας πολιτικός διάλογος με τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Και εγώ ο ίδιος ε, και από πλευρά του κυρίου Βούτσιτς που πήγε στο Κωσυφοπέδιο και συζήτησε με τους Σέρβους στο βορρά του Κωσυφοπεδίου, στόχος μας είναι, κοινή μας προσπάθεια είναι να καταφέρουμε να συμμετάσχουν οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου στο μεγαλύτερο δυνατό εφικτό στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Όπως σας είναι γνωστό, το σχέδιο ε, εφαρμογής προβλέπει και την ε, τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές όσον αφορά την ε, δικαστική εξουσία και την αστυνομική, τις αστυνομικές αρχές που θα πρέπει με ε, τα, τις αλλαγές και τα, το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα υλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Έχουμε και βραχυπρόθεσμα μέχρι τις 28 Ιουνίου συγκεκριμένο έργο που πρέπει να επιτελεστεί. Όμως η διαδικασία αυτή δεν θα μπορέσει μόνο μέχρι τότε να υλοποιηθεί πλήρως. Αυτό που μετρά φυσικά είναι ότι όλοι θα πρέπει να πιστούν ότι δεν είναι θέμα εξαγοράς χρόνου ή κάποιων προσχηματικών κινήσεων ε, προς όφελος κάποιων. Όχι. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αυθεντική προσπάθεια. Θέλω να τονίσω τον θετικό ρόλο της κυρίας Άστον και θέλω να την ευχαριστήσω για έναν πολύ θετικό ρόλο που διαδραμάτισε σε σχέση με τις ε, ε, συζητήσεις που είχαμε. Όταν η Hillary Κλίντον και η Λέδη Άστον προσήλθαν στο Βελιγράδι και ο κύριος Νίκολιτς και εγώ είχαμε επαφές και συζητήσεις μαζί τους. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου και οι δύο εκπρόσωποι εντυπωσιάστηκαν ότι εγώ στη συνέντευξη τύπου είπα ακριβώς αυτά τα οποία είχα αναφέρει προηγούμενα. Διότι είναι συνηθισμένο κάποιοι να λένε κάτι σε κάποια συνεδρίαση και μετά να αναφέρουν κάτι άλλο σε συνέντευξη τύπου. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι δεδομένο που αξιολογήθηκε θετικά από τις δύο εκπροσώπους. Μπορούμε λοιπόν ε, με θετικό τρόπο να εκφράζουμε τις απόψεις μας και άμεσα να λέμε τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και τι όχι. Και για πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, ε, ζητήσατε να μάθετε για την αναδιάρθρωση της κυβέρνησης και της προσπάθειάς μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί εν ευθέτω χρόνο δεδομένης της περίοδου που ε, αναμένει συγκεκριμένη δράση από εμάς ε, στο άμεσο μέλλον, η Σερβία χρειάζεται ένα πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας για να συνεχίσει την πορεία της, ε, άσχετα από το αν κάποιοι παραμείνουν υπουργοί σε μια κυβέρνηση ή όχι. Δεν γνωρίζουμε όμως ακριβώς ποιος θα είναι ή ποιος θα έχει συγκεκριμένο αξίωμα. Αναφέρθηκε από τον συνάδελφο το θέμα των αρχείων της πρώην Ιουγκοσλαβίας δεν είμαι τόσο νέος, είμαι 47 ετών και δεν πιστεύω ότι εγώ αποτελώ μέρος ή τμήμα αυτών των αρχείων, παλαιότερων δηλαδή αυτών αρχείων της πρώην Ιουγκοσλαβίας θα μπορούσαμε όλα να τα εξετάσουμε όσα δεν αντιβαίνουν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ε, ή και της ε, ε, περιοχής μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με αυτή την πτυχή αυτής της συμφωνίας. Και όσον αφορά τη σχέση μας με τις όμορες χώρες και τις κυβερνήσεις τους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας θα πρέπει να έχουμε επαφές με τις πρωτεύουσες αυτές, με τις χώρες αυτές έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες είναι κοντά μας γεωγραφικά αλλά δεν είναι τόσο κοντά μας όσον αφορά την, ε, την συγκοινωνία και τις, ε, ε, την οδική και άλλη σύνδεση μαζί τους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί ο διάδρομος 10, Corridor 10, ο διάδρομος 11 ώστε να συνδεθούμε με τις χώρες αυτές, να συνδεθούμε με την Ρουμανία και το Σαράγεβο. Δεν έχουμε, βλέπετε, αυτοκινητόδρομο μέχρι τώρα. Όμως στην συνεδρίαση τίνεται να υπάρξει ένας αυτοκινητόδρομος μεταξύ Πρίστινα και Νίσ, μια πόλη στη Νότια Σερβία και να συνεχιστεί από εκεί προς την Ουγγαρία και προς την Βουλγαρία. Πολλά βαριά οχήματα φορτηγά κυκλοφορούν σε αυτή την περιοχή και οι δρόμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ε, αντιμετωπίζουμε δύσκολα θέματα ε, και εξετάζουμε τα θέματα αυτά και με την κυρία Άστον. Δεν υπήρξε συμφωνία για το θέμα του ε, αυτοκινητοδρόμου. Υπήρξε πρόταση να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση ή τοποθέτηση μέχρι τώρα. Δεν έχει επιτευχθεί λοιπόν συμφωνία με την ε, κυρία Άστον ε, Παρτών. Δεν μπορούμε απλά να αναμένουμε χρήματα, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι απλά, αλλά είναι πρωτοβουλίες από την κυβέρνησή μας και η ε, κυβέρνηση συνασπισμού υποστηρίζει πλήρως ε, αυτές τις πρωτοβουλίες. Και όσον αφορά την ολοκλήρωση, την ε, ένταξη των αστυνομικών σε άλλες νέες δομές, η αρχή νομίζω είναι σαφής και έχει εξεταστεί και όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί δεόντως ώστε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ε, παραβεί τον, λόγο, τον νόμο θα πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν στα νέα θεσμικά όργανα, στους νέους θεσμούς. Άλλοι οι οποίοι συμμετείχαν ε, σε κάποια εγκληματική πράξη δεν μπορούν να το πράξουν αυτό και δεν μπορούν να αποτελέσουν προσωπικό αυτών των ε, ε, μονάδων στο μέλλον και οικονομικά μέτρα είναι θεμελιώδους σημασίας ε, για την Σερβία. Αναλύθηκαν πρωτοβουλίες και αφενό ε, πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι σημαντικά. Από την άλλη πλευρά πρέπει να προσελκύσουμε το δυνατόν το υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στη χώρα μας και να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και να σημειώσουμε πρόοδο αν δεν αναπτύξουμε τη Σερβία και όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν και υπό τους όρους ε, δαπανών για την, το αναγκαίο διοικητικό πλαίσιο πρέπει να υπάρξει να, η μείωση μισθών και συντάξεων είναι κάτι δυσχερέστατο διότι ένας ε, μέσος μισθός στο Βελιγράδι είναι 365 ευρώ και η κατάσταση με τις αλλαγές που σημειώνονται και οι συντάξεις που είναι το ίμιστο των ε, μισθών δείχνουν σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε πάρα πολύ δύσκολο να πει κανεί θα μειωθούν περαιτέρω και οι μισθοί και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο και οι συντάξει. Έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να κινηθούν προς μια κατεύθυνση ε, κοινωνικής ανάπτυξης ε, κατά 2% πιστεύουμε. Αυτό όμως ε, δεν επαρκεί. Θα έπρεπε να είναι 5% το ποσοστό ανάπτυξης που θα σημειωθεί κατά το τέλος της περίοδου, ώστε να υπάρχει ένα ορατό πλαίσιο, ευδιάκριτο πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης που θα επιτευχθεί. Αυτά που έγιναν κατά το 2012 ήταν κάτι που υποστηρίχθηκε και ομόφωνα, ομόθυμα από πλευράς της ε, κυβέρνησης ε, και ε, της συμπολίτευσης και πρέπει εδώ να αναφέρω ότι πολλά σε σχέση με την συμφωνία δεν, δεν υποστήριξαν απλά και μόνο τα μέρη αυτής της συμφωνίας αλλά την γενικότερη κατεύθυνση, την ανάγκη να κινηθεί προς τα εμπρός, να σημειώσει πρόοδο η Σερβία. Δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε τον ρόλο μας όσον αφορά αυτή την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί. Διότι αυτά που επετέφθησαν είναι κατά κύριο λόγο θετικά για τη Σερβία και τους πολίτες της Σερβίας. Είναι ηρωνικό, είναι μια πολιτική ηρωνία. Το μόνο κόμμα στο κοινοβούλιο που αντιτίθεται είναι το κόμμα του Βόισλαβ Κοστούνιτσα εκείνου δηλαδή που με άλλα λόγια ήταν εκείνος ε, που ε, υπέστη αυτή την ε, ήττα. Δίνεται όμως σε κάθε κόμμα η δυνατότητα να έχει τη δική, της, τη δική του θέση. Θα ήθελα να ζητήσω σε σχέση με αυτά τα θέματα να σας ζητήσω να, συμπεριληφθεί, να συμπεριληφθούν και οι δικές μας, ε, τα δικά μας κόμματα, τη δική μας Βουλής σε αυτό το ε, γίγνεσθε, το ευρύτερο ε, πολιτικό γίγνεσθε, να μπορέσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε με αυτές τις αξίες στις ευρύτερες προσπάθειες. Το δικό μου κόμμα έχει κάποια προβλήματα με τα θέματα στην ένταξη στην ε, σοσιαλδημοκρατική ε, ομάδα ή τη σοσιαλιστική ομάδα. Και προβλήματα τα οποία συναρτώνται με τις εσωτερικές ε, πολιτικές που ακολουθούμε. Ε, μία άλλη ομάδα που δεν βρίσκεται στην εξουσία όμως ε, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι κάτι το αποκλειστικό ε, και το κόμμα του κυρίου Βούτσιτς, το Σοσιαλιστικό Προοδευτικό Κόμμα το να μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως για παράδειγμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αυτονομία της Βορβοδίνας, δεν έχουμε κάποιο, κάποια πρόθεση να περιοριστεί η αυτονομία αυτή όσον αφορά το καταστατικό της. Δεν είναι δυνατόν όμως να είναι κράτος εν κράτη και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όλοι είπαν ότι η σερβική κοινότητα στο Κωσυφοπέδιο δεν μπορεί να είναι μια ρεπούμπλικα σέρβσκα και έτσι λοιπόν η Σερβία δεν είναι δυνατόν να πει ότι ορίστε η Βοηβοδίνα λοιπόν ας έχει κρατικές ε, ε, προοπτικές και κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν πρέπει αυτά να αντιβαίνουν λοιπόν τα ε, σερβικά συμφέροντα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ακολουθηθεί η πολιτική μιας πολιτικής αυτονομίας όμως μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης πραγμάτων της Σερβίας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να εξευρεθούν σαφείς κανόνες και κανονισμοί για τέτοιου είδους προοπτικές. Δεν είναι κατά της ένταξης του κοσυφοπεδίου στα ε, περιφερειακά φόρα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν τα πράγματα να ολοκληρωθούν ε, με τη συμφωνία την οποία συνάψαμε, πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να πάρουν σάρκα και οστά. Τώρα θα πρέπει να βρούμε ένα επαρκές ικανοποιητικό πλαίσιο που θα δώσει την δυνατότητα αυτής της συμμετοχής. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να, με κάθε σοβαρότητα να προσεγγίσουμε την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων και να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Να μην τα αντιμετωπίσουμε ε, με την ε, ε, ακύρωση ή απαγόρευση τέτοιων πρωτοβουλειών. Είναι θέμα αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Δεν έχει κανένα συμφέρον η Σερβία, για παράδειγμα, αν έχουμε έρθει σε επαφή με τον Θάτσι δέκα φορές για παράδειγμα και με την ε, υποστήριξη της κυρίας Άστον δεν θα ήταν λογικό εμείς ε, να είχαμε ε, συζητήσεις με τους εκπροσώπους της Πρίστινα σε άλλα φόρα, σε άλλα επίπεδα και θα πρέπει να δούμε σε ποια φορά, σε ποια θεσμικά όργανα θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε το θέμα αυτό να διευθετηθεί στην ημερήσια διάταξη και να πάψει να αποτελεί πρόβλημα. Ενδιαφερόμαστε στην περιφερειακή ασφάλεια. Θέλουμε να έχουμε στενές σχέσεις με όλους ε, στην ε, ε, περιοχή μας και με την Ρουμανία θα έχουμε ανοιχτές ε, ε, ολοκληρωμένες επαφές ε, καθώς επίσης και με τα θέματα τα οποία εφίστανται στην Ανατολική Σερβία. Η Ρουμανία και η Σερβία είναι μεγάλοι φίλοι, όμως η Ρουμανία ακόμα και όταν η Γερμανία μας έδωσε το πράσινο φως, η Ρουμανία δημιούργησε, έθεσε το θέμα όταν μας αναγνωρίστηκε το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τέτοιου είδους προβλήματα να τα αντιμετωπίζουμε ώστε να διευθετούνται με τον ευθετότερο τρόπο. Όσον αφορά την Μακεδονία, λέει ο μιλητή, θα έχουμε μια συνάντηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Επιθυμούμε να έχουμε στενότατε σχέσει, όπω επίση και με το Μαυροβούνιο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε την καθυστέρηση και να ξεπεράσουμε και την απόσταση που μα χωρίζει από χώρε που ε, έχουν κάποιε διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ευχόμαστε τίποτα το αρνητικό ει βάρο αυτών των χωρών. Ευχόμαστε μόνο κάτι το πολύ θετικό υπέρ τη και δεν έχουμε κάποιες προκαταλήψεις ή ιδεολειψίες όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις ε, στην ευρύτερη περιοχή λόγω του ότι είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη χώρα και έχουμε σχέσεις φυσικά με την Τουρκία. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε υπέρ η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή να παραμείνει, ας το πω έτσι, στην διακριτική ευχέρεια κάποιων ε, τρίτων. Και προτού τοποθετηθώ στο θέμα των σχέσεών μας με την Τουρκία ή τη Ρωσία, αν κάποιος δεν είναι παρόν και δεν δραστηριοποιείται στην περιοχή μας, κάποιος άλλος μπορεί να καταλάβει αυτό το χώρο. Η Σερβία έχει μεγάλο, επί μεγάλο χρονικό διάστημα φιλικές σχέσεις με την Ρωσία και είναι όμως και προς το συμφέρον της Σερβίας να έχει εταίρους ε, και στην Δύση και όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Δυτική Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και αναζητούμε τέτοιου είδους ε, εταιρικές σχέσεις ε, Γι' αυτό έχουμε και συμφωνίες με τη Γαλλία και την Ιταλία επιστρατηγικού χαρακτήρα συμφωνιών και εταιρικών σχέσεων και με την Κίνα και τη Ρωσία επίσης. Να μην έχετε καμιά αμφιβολία. Η Ρωσική Ομοσπονδία με τη Σερβία σκοπεύει να αναπτύξει με ειρηνικό τρόπο τις οικονομικές και οποιασδήποτε άλλες σχέσεις χωρίς οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Το αντίθετο κιόλας συμβαίνει. Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακόμα καλύτερες οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία από τη ίδια η Σερβία σήμερα. Και τέλος, μια και αναφέρατε την Τουρκία, επ' αυτού θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο όρος Βαλκάνια, λένε κάποιοι κάτι άλλο, όμως Βαλκάνια είναι το όνομα μιας οροσυράς Μπαλκάν στην Βουλγαρία και ουσιαστικά πρόκειται για δύο τουρκικές λέξεις Μπαλκ και Καν. Το ένα σημαίνει αίμα, το άλλο μέλι, λέει ο κύριος Ντάτσιτς. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πιούμε ένα ποτήρι μελιού, ένα ποτήρι μέλι, γλυκό ποτήρι και όχι αίμα. Και όταν η κυβέρνηση της Σερβίας δημιουργήθηκε υπήρχαν πολλά διλήμματα και προβλήματα σε σχέση με αυτό. Ο, αισθάνθηκα όμως ότι μια και τίποτα δεν αναμενόταν που να ήταν θετικό από τη Σερβία και οτιδήποτε ε, κάναμε θα έπαιρνε ε, ένα ε, μεγάλο συν, θα εξετιμά ίσως θετικά. Τώρα υπάρχουν και ε, άλλες προοπτικές αναμένουν πολλά περισσότερα από τη Σερβία με τις προσδοκίες τους. Ε, λες και είμαστε παντοδύναμοι. Και τώρα η δουλειά μας δυσχεραίνεται ιδιαίτερα επειδή πρέπει να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε την ε, συνέχιση της πορείας μας προς μια νέα πολιτική, προς μια νέα ε, εποχή κυρίως επειδή οι πολίτες μας, οι ίδιοι οι πολίτες της Σερβίας το χρειάζονται αυτό και σας ζητώ απευθύνω έκκληση να μας βοηθήσετε, να συνδράμετε την Σερβία, να δώσετε την έγκριση στη Σερβία για έναρξη διαπραγματεύσεων προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικότατο μήνυμα για την ε, κατάσταση της Σερβίας της ίδιας αλλά και την θέση της ε, στα Βαλκάνια. Είσαστε ευπρόσδεκτοι, μπορείτε να, να έρθετε στη Σερβία όποτε επιθυμείτε και σίγουρα δεν θα ξεχάσετε αυτή την επίσκεψή σας στη χώρα μας γιατί είμαστε τόσο φιλόξενος λαός. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ για όλες σας τις απαντήσεις, για τα καλά νέα που μας φέρατε, για την ευγενική σας πρόσκληση. Είναι αποδεκτή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως και γεια σας. Thank you. We are uh,